Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Έχουμε λίγο χρόνο και πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης ε, είχαμε και την τύχη να έχουμε μια προσκεκλημένη ακριβέστατη. Για την έγκριση της ημερήσιας διάταξης ε, θα ήθελα να σας θυμίσω, ίσως βέβαια να το ξέρετε συνάδελφοι, ότι ο, ο Κροάτης Υπουργός Εξωτερικών που θα έπρεπε να έρθει σήμερα δεν θα έρθει διότι σήμερα στην Στοκχόλμη υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας για να λυθεί αυτή η ε, διαμάχη ε, σχετικά με τα σύνορα. Λοιπόν, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η απουσία του. Θα την αντισταθμίσουμε όμως με την παρουσία του δόκτωρα Βλάντιμιρ Ντρόπνιακ ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Κροατίας για την προσχώρηση. Η ανταλλαγή απόψεων με τον στρατηγό Μοριγιό για αύριο το απόγευμα έχει ακυρωθεί και αυτό λόγω της απεργίας των τρένων στο Βέλγιο και στη Γαλλία και θα γίνει η συνάντηση αυτή στις 10 Νοεμβρίου στις 4 όπου πέρα του κυρίου, του πρώην συναδέλφου μας ε, Μοριγιό θα είναι και ο συνάδελφος Μπέρμαν ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων Παρατηρητών για τις προεδρικές εκλογές ε, <clears throat> στο Αφγανιστάν που ακυρώθηκαν λόγω της απόσυρσης από, την εκλογική μάχη του Αμπδουλά Αμπδουλά Αυτά για τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Για να μην καθυστερούμε παραπάνω την φιλοξενούμενη μας, θα προχωρήσω στις ανακοινώσεις της Προεδρίας μετά αφού χαιρετήσω βέβαια για τα λίγα λεπτά που θα είναι παρόντες εδώ μία αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας της οποίας προεδρεύει η πρόεδρος του Ισλανδικού Κοινοβουλίου, η κυρία Ντότερ και συνοδεύεται από τον πρέσβη Τζόνσον. Αγαπητοί Υπουργέ και συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου χαρά που είστε μαζί μας σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν ορισμένες αποφάσεις από το Συμβούλιο που ενδιαφέρουν άμεσα στην Επιτροπή μας και που θα πρέπει να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα. Αυτά ως, τα δίνω ως γενικές εξαγγελίες, μετά θα τα αναλύσουμε όλα αυτά τα σημεία. Οι οδηγίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, επιτρέψτε μου να πω ότι το Συμβούλιο καθόρισε τη γραμμή του Καθόρισε λοιπόν την ε, γραμμή του βασιζόμενο και στη γνωμοδότηση που εμείς ε, ε, εκπονήσαμε ως κοινοβούλιο. Διότι εμείς δίνουμε και την κατεύθυνση στον προϋπολογισμό για το πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι υπηρεσίες. Εμείς αισθανθήκαμε σχετικά παραμερισμένοι στις αρμοδιότητές μας ως κοινοβούλιο. Αλλά ελπίζουμε ότι με τον προπολογισμό θα τα αναπληρώσουμε. Λοιπόν, υπογράφηκε και η Συμφωνία Συνεργασίας με τη Συρία που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια να σας θυμίσω ότι θα πρέπει να συνενέσει σχετικά και η Επιτροπή μας για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, ε, αποφασίστηκε μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, που πέρα από την ε, στρατιωτική παρουσία θέτει σε μια πρώτη γραμμή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα αστικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών. και γενικότερα τους πολιτικούς ε, στόχους που πρέπει να προσεγγιστούν και όχι μόνο τη στρατιωτική παρουσία. Θα μπορούσαμε να καθορίσουμε αυτή τη στρατηγική όχι ως μία στρατηγική εξόδου όπως θέλησαν να την ορίσουν πολλοί, αλλά ε, μία στρατηγική προοπτικών όπως το είχε πει και ο κύριος Σολάν εδώ ούτως ώστε στην νέα δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Αφγανιστάν να δοθεί ένα σχήμα ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στη σύσταση μιας κοινωνίας δημοκρατικής και ευήμερης. Εμείς έχουμε λοιπόν τώρα μια ε, νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση και έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ε, με όλη την ε, συνεργατικότητα την οποία γέννη επιδεικνύουμε. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε κυρία Υπουργέ. Ε, θέλω να σας πω ότι... Σας τα λέω τώρα για να μην θυμώσετε μετά αλλά να σας θυμίσω τον αντιπαθητικό μου ρόλο ως πρόεδρο που πρέπει να ρυθμίζω τις χρονικές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Μετά από 7 χρόνια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επανέρχομαι, είναι, βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά μου, δέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρόσκληση. Είμαι έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις, αλλά βρίσκομαι εδώ για να σας αναφέρω το τι συνέβη τη Δευτέρα και την Τρίτη στην, στο, ε, συνεδρίαση εξωτερικών υποθέσεων. Το πρώτο τμήμα αφορούσε στα συμπεράσματα ως αποτέλεσμα των συζητήσεων στη διάσκεψη κορυφής που ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν στα βασικά θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Αρχίσαμε με το δείπνο, Δευτέρα βράδυ. Ιράν και Δυτικά Βαλκάνια ήταν το θέμα της συζήτησης. Το Ιράν βρίσκεται στη μεσχεδιάταξη διάταξη διότι όπως όλοι γνωρίζετε η κατάσταση είναι ταραχώδης μετά το καλοκαίρι με ευρύτατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έλλειψη βούλησης από πλευράς καθεστώτος να συνεργαστεί επικοδομητικά με τη διεθνή κοινότητα. Η Προεδρία έχει, έχει δημοσιεύσει σειρά δηλώσεων ε, σχετικά με τις καταθέσεις των διαφωνούντων και θανατικές ποινές. Μας απασχολούν οι μαζικές δίκες μετά από διαδηλώσεις και η μη εφαρμογή διεθνών ε, προτύπων που το Ιράν έχει προσυπογράψει. Επίσης παραβιάζει συνταγματικές αρχές και διατάξεις. Σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία ε, παραμένουν, ε, παραμένουν παραμένουμε ενιαίοι ε, και συμπαγείς. Θέλουμε να δείξουμε ότι αν το Ιράν ε, αντιληφθεί ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος, δρόμος συνεργασίας παρά αντιπαράθεσης, είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε. Τον Οκτώβριο, πριν από λίγες εβδομάδες, οι πολιτικοί διευθυντές από του 3 ε, συν 1 συναντήθηκαν με τον κύριο Τζαλίλη, τον επικεφαλής διαπραγματευτή. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά από 14 ε, μήνες και μετά την αποκάλυψη μιας νέας μονάδας για εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν. Η συνάντηση δεν είχε πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα ε, μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά το Ιράν δέχθηκε να ανοίξει τις εγκαταστάσεις προς την EIA για έλεγχο και επίσης είναι πρόθυμο να συνεργαστεί για εξαγωγές ουρανίου ώστε να ε, ε, ε, εμπλουτιστούν έτσι περαιτέρω. Μέχρι στιγμής βέβαια στα βασικά ερωτήματα έχουμε πάρει γενικές απαντήσεις, ενώ η δεύτερη συνάντηση του Οκτωβρίου δεν υλοποιήθηκε. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων η ε, υπουργοί οι υπουργοί αναφέρθηκαν στα επιμέρους θέματά τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επαφές με άλλες χώρες. Επίσης, επανέλαβαν την προσέγγιση, την διτής κατεύθυντης προσέγγιση και επίσης την επιμονή για αποκλειστικά ειρηνική χρήση ε, το, της πυρηνικής ενέργειας. Οι υπουργοί συμφ Συμφώνησαν επίση ότι υπάρχει δυσκολία να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της τάση του Ιράν. Πολλοί υπουργοί δεν ήταν υπερβολικά αισιόδοξοι σχετικά με το μέλλον και υπογράμμισαν ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος μέχρι το τέλος του έτους και κάποιοι ισχυρίζονται ότι η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν παραβιάζοντας τα ψηφίσματα του ΟΗΕ η συνέχιση αυτή μπορεί να καταλήξει σε ε, επιπρόσθετες κυρώσεις. Κάποιοι άλλοι υπουργοί είπαν ότι για να είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις θα πρέπει να αποφασιστούν από τον ΟΗΕ και συμφωνήθηκε ότι χρειάζονται στοιχεία και δεδομένα για να ε, αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των πιθανών κυρώσεων. Έγινε επίση μια σύντομη συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια και κυρίω βοσνια Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου η Προεδρία έδωσε τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου συνομιλιών που έλαβαν χώρα μεταξύ ΕΕ και των ηγετών της Βοσνίας στο Καμπούντι έξω από το Σαράγεβο στις 21 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτιών ήταν ο Μπίλτ, ο κ. Στάιμπεκ, ο Ρίρ και ο Γενικός Διευθυντής κ. Κούπερ και επτά διαφορετικοί ηγέτες από βυθιακής πλευράς. Το Συμβούλιο καλωσόρισε την πρωτοβουλία υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα της Βοσνίας και θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες για μεταρρυθμίσεις ευρείας κλίμακος. Η συνάντηση αυτή δεν κατέληξε σε ουσιαστικά αποτελέσματα διότι οι ηγέτες της Βοσνίας ε, κράτησαν μαξιμαλιστικές θέσεις και δεν υπάρχει διάθεση για ε, υποχωρήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια συγκρατημένη αισιοδοξία ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος. Στις προσεχείς εβδομάδες θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη συνέχιση της διαδικασίας, να ακούσουμε τις διάφορες πλευρές και να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την λειτουργικότητα του κράτους. Τα μέρη θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να περιοριστούν στο απόλυτο ελάχιστο. Ε, πρέπει να προχωρήσουν και μόνο αν υπάρξει μεταμόρφωση μετασχηματισμός μάλλον και να διαπιστωθεί αυτό από το γραφείο του ανώτατου εκπροσώπου, μόνο τότε θα μπορέσει να υποβάλει ε, την αίτηση η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πολύ σύντομα συζητήσαμε και το ζήτημα της Αλβανίας. Ε, για διαδικαστικούς λόγους δεν ήταν δυνατόν να σταλεί η αίτηση για γνωμοδότηση. Ελπίζουμε όμως ότι τούτο θα γίνει το Νοέμβριο. Το επόμενο πρωί ε, ασχοληθήκαμε με το θέμα της Μέσης Ανατολής, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή όπου η ερνευτική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, εντάσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ε, άσχημη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Δεν υπάρχουν ορατά αποτελέσματα, η παριστινιακή πλευρά παραμένει εγκλωβισμένη στο διχασβό. Ε, αναφέρθηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξει μια γενική συζήτηση έτσι με αυθόρμητες παρεμβάσεις για το τι μπορεί να γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε η συζήτηση με τον κύριο Σολάνα, ο οποίος έκανε μια περιγραφή της τελευταίας επισκεψής του στην περιοχή και υπογράμμισε το, ε- τον επίγοντα χαρακτήρα στην να αρχίσουν διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος του έτους. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να υποστηριχθεί το σχέδιο Φαγιάτα σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πάντα θα πρέπει να είναι πολύ σαφής ευθύς εξ αρχής για το στόχο ε, των δύο κρατών ε, τη βάση των αποφάσεων του 2006. Επίσης ε, υποστηρίζουμε την ε, πρωτοβουλία Ομπάμα και τις δεσμεύσεις από αραβικής πλευράς υπέρ ε, επίσης της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή πλευρά και τον πρόεδρο Αμπάσα. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην οικοδόμηση του κράτους, στην ασφάλεια, τους πρόσφυγες ενώ πολλοί υπουργοί διατύπωσαν ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τόνισαν ε, την ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση στην περιοχή. Επίσης ε, θα πρέπει να υποστηριχθεί η διαπαλαιστινιακή συμφιλίωση και οι προσπάθειες ε, παρέμβασης από την Αίγυπτο. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να σταματήσει αυτός ο διχασμός μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας και θα αποκατασταθεί η ενότητα ε, των Παλαιστινίων εν ώψη ενός μελλοντικού ενιαίου κράτους. Συζητήθηκε και το Αφγανιστάν, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα να πω. Τότε θεωρήσαμε ότι θα υπάρξει δεύτερος γύρος ε, εκλογών, τώρα γνωρίζουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, ωστόσο το Συμβούλιο υιοθέτησε, όπως είπα, είπε και ο Πρόεδρος, τα συμπεράσματα αναφέρθηκε στη στρατηγική για περαιτέρω υποστήριξη από Ευρωπαϊκή Ένωση προ το Αφγανιστάν και Πακιστάν. Αυτά είναι σημαντικά, θεωρούμε, και θα καθοδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προβλέψιμο μέλλον. Και ε, επίση υποβλήθηκαν δύο ε, μπλε βιβλία στο Συμβούλιο για την κατάσταση του Πακιστάν και του Αφγανιστάν συνολικά πάνω από ένα δις ευρώ, σε πάνω από ένα δις ευρώ ανέρχεται η βοήθεια προς το Αφγανιστάν. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών, να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί όπου υπάρχει προστιθέμενη αξία. Ε, οικοδόμηση του κράτους, καλλιδιακή κυβέρνηση, κράτο δικαίου. Η σημασία ενίσχυσης της ε, EUPOL, επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, οργανώνει μια νέα αποστολή 100 παρατηρητών, επίσης ε, υπογραμμίζεται η ανάγκη για ανάληψη της ευθύνης από αφγανικής πλευράς. Συζητήσαμε την διοργάνωση μιας διάσκεψης μετά την συγκρότηση της κυβέρνησης και το συνέδριο κατά προτίμηση θα διεξαχθεί στην Καμπούλ. Και βέβαια η κατάρτιση της ατζέντα είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Πακιστάν. Οι υπουργοί αναφέρθηκαν στην επιδεινούμενη κατάσταση και την ανάγκη υποστήριξης ε, της κυβέρνησης να ε, καταπολεμήσει τους ένοπλους ε, κατάσταση στη Σριλάνκα. Η εσωτερική διαμάχη σταμάτησε τον Μάιο, αλλά ακόμα υπάρχουν σοβαρά ανθρωπιστικά προβλήματα. Πάνω από 250.000 εσωτερικώς εκτοπισμόνι βρίσκονται σε εγκαταστάσεις και στρατόπεδα και δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτούς. Το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα για να καλέσει την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρόοδος προς την επίλυση των συνεπειών της σύγκρουσης ε, είναι βραδύτατες και η όλη διαδικασία συμβιλίωσης επιβραδύνεται. Όλες οι κοινότητες της Ρελάνκα θα πρέπει να εμπλακούν. Υπάρχουν σοβαρές ε, εκθέσει σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων για απαγωγές, βιασμούς και άλλες βιότητες. Το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του επαναλαμβάνει το, την έκκληση για διακοπή των βιαιοτήτων και για αποκατάσταση μιας ε, σταθερότητας που είναι απολύτως απαραίτητη για τη συμβιλίωση κυβέρνηση της ε, Σρι Λάνκα ανέφερε ότι μεγαλύτερος αριθμός των εκτοπιστέντων θα επανεγκατασταθεί ε, στις περιοχές από όπου έφυγαν και αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες. Επίσης οι Υπουργοί ε, δήλωσαν ότι χρειάζεται ενίσχυση, υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης της κυβέρνησης. Μολδαβία. Ο κύριος Καρλ Μπίλτ ήταν επικεφαλής της ε, Τρόικα ε, στην επίσκεψή της στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Η Μολδαβία αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κατάσταση και θα πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Έχει μια νέα κυβέρνηση, συμμαχία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, επικεφαλής ο κύριος Μιλάτ, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι πρώτη προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει. Μια νέα συμφωνία είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Η Μολδαβία αποτελεί μέρος του προγράμματος ε, ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τρόπους επιτάχυνσης χρηματοδοτικής υποστήριξης ώστε να συμπληρωθούν τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ως προς την υπερνηστερία, τη σύγκρουση εκεί, Υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις 2 συν 1 και στη συζήτηση που ακολούθησε οι Υπουργοί τόνισαν ε, την ανάγκη να ε, υποστηριχθεί η Μολδαβία τώρα που υπάρχει μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στη χώρα. Αυτά ήταν κύριε Πρόεδρε τα βασικά θέματα συζήτησης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν ιδιαίτερα ολοκληρωμένοι και σύντομοι. Ξαναλέω ένα μόνο λεπτό τοποθετήσεις. Μία μόνη ερώτηση. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε καλωσορίζουμε αγαπητοί συνάδελφε Μάλστρομ Ξέρουμε ότι έχεις αναλάβει όμως άλλες ευθύνες. Θα ήθελα να ξέρω. Ποιο είναι το θεσμικό χρόνο χρονοδιάγραμμα για το έκτακτο συμβούλιο μετά την υπογραφή φυσικά της συνθήκης από τον πρόεδρο της Τσεχίας το χρονοδιάγραμμα δηλαδή για το διορισμό των επιτρόπων και την παρουσίασή τους εκεί. Θα ήθελα να ξέρω τώρα για το δεύτερο γύρο των εκλογών στο Αφγανιστάν και υπό το φως των συμπερασμάτων ε, του Συμβουλίου γιατί άλλαξε η... η εικόνα που έχουμε για τη Συριανή κυβέρνηση για να υπογραφεί δηλαδή η συμφωνία. Τι έχει αλλάξει. Και τι γίνεται με, τις, ε, την Ονδούρας. Λοιπόν, τώρα με, με τις αλλαγές που μεσολάβησαν, τι θα γίνει με τις συμφωνίες συνεργασίας. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Ο κύριος Κρέις Δόρφρερ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, για το Αφγανιστάν. Ο νέος υπουργός ε, αμήνης ε, Φον Κούτας στη Γερμανία χαρακτήρισε το Αφγανιστάν ως ε, εμπόλεμη περιοχή. Ξέρουμε στο διεθνές δίκαιο τι σημαίνει πόλεμο, Πόλεμο σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται παραδείγματος χάρη με τους του πολέμου. Εσείς πώς το βλέπετε το θέμα, μπορείτε να συμφωνήσετε με την εκτίμηση αυτή του κυρίου Τζουγκούτενμπερκ και τι γίνεται με το Αφγανιστάν, όπου όλοι προσπαθούν τώρα να φύγουν πάλι. Εγώ δεν βλέπω ε, ε, βραχυπρόθεσμα συγγνώμη, καμία ευκαιρία κάτι τέτοιο, ούτε μεσοπρόθεσμα. Θα διαρκέσει πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα τι θα γίνει εκεί. Και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο απομακρυσμένο το να χαρακτηρίσουμε ότι είναι μια εμπόλια. E Ευχαριστώ κύριε Ντόρφλερ. Ο κύριος Βότσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρω μπορώ να χαιρετήσω την Προεδρεύουσα. Μα έλειψε πολύ και είναι ευχαρίστηση μέσα να την έχουμε εδώ. Ήθελα να τη συγχαρώ επίση για μια συμβιδική Προεδρία που όσο πάει και πιο πολλά υποσχόμενη δείχνει. Η Προεδρεύουσα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η συνθήκη της αγώνας θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, ότι η Προεδρία θα οργανώσει μια έκτακτη διάσκεψη κορυφής την επόμενη εβδομάδα και ότι ο Τόνι Μπλερ δεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Συμβουλίου. Θα ήθελε επίσης να μας ε, πει γιατί δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση της ε, καταπολέμησης ε, των ε, κλιματολογικών αλλαγών στο Συμβούλιο την περισμένη εβδομάδα και επίσης γιατί το Ιράν θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ κύριε Βότσον. Η κυρία Λούνατσεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Προεδρεύουσα, τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η μία για το κοσυφοπαίδιο. Και πώς φαντάζεστε ότι θα αναπτυχθεί η κατάσταση στο Συμβούλιο την επόμενη σύνοδο όσον αφορά την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων διαβατηρίου για το ψυχοπαίδιο μια έκθεση πρόοδου του κυρίου Ρεν λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος για τις θεωρήσεις με στόχο την απελευθέρωση. Βλέπετε και εσείς τα πράγματα υπό την ίδια σκοπιά. Δεύτερον, η έκθεση πρόοδου αναφέρει επίσης ότι η Μακεδονία ή μάλλον με τη Φύρο θα πρέπει να ξεκινήσουν. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, κυρία Λούνασεκ. Το λόγο έχει η συνάδελφο Άτκινς για ένα λεπτό. Ο συνάδελφο. Πολύ σύντομα, πρόεδρε. Σήμερα που σκοτώθηκαν άλλοι πέντε Βρετανοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν, δεν ξέρω αν η Προεδρεύουσα μπορεί να μας πει κάτι ε, όσον αφορά την αποστολή από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ στρατιωτών στο Αφγανιστάν για να υποστηρίξουν τους Αμερικανούς και ε, Βρετανούς στρατιώτες που βρίσκουν εκεί. Θεωρείται επίσης ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα επίλυση των προβλημάτων διαφθοράς που υπάρχουν στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Κάτι όπως αυτό που είπε ο πρόεδρος Ομπάμα για μια δράση έξι μηνών που δεν πρέπει να παραμείνει λόγια. Και κάτι ακόμα. Συζητήθηκε τίποτα και μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά όσον αφορά τα προβλήματα των Παλαιστινίων στην Γάζα, υποστήριξη υποδομή ε, μεταφορές, δημόσια υγεία και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ κύριε Άτκινς. Συνάδελφος Μέιερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Η προσυμφωνία μεταξύ της ε, πραξικοπηματικής κυβέρνησης και της νόμιμης κυβέρνησης στην Ονδούρας ε, έγινε ε, μετά από την συνεδρίαση του Συμβουλίου. Αλλά θα ήθελα να ξέρω, επειδή ένα από τα σημεία κλειδί αυτής της συμφωνίας είναι η αποκατάσταση του Προέδρου Θελάια από το Κογκρέσο της Ονδούρας, θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα γίνει με τη Συμφωνία Συνεργασία. Ξέρω ότι ο ΟΗΕ παρακολουθεί για την απόλυτη πλήρωση των όρων της συμφωνίας. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Υπουργέ, σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί ο κύριος Θελάγια, τι θα κάνει το Συμβούλιο, θα ακολουθήσει την γραμμή του ΟΗΕ να μην αναγνωρίσει δηλαδή την πληξικοποιηματική κυβέρνηση του Μισελέ. Ευχαριστώ κύριε Μέιερ. Ο κύριος Κασουλίδης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. Πρώτον, θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό εάν μπορεί να αξιολογήσει το ρόλο της Σερβίας στις στις προσπάθειες της ΕΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, Βοσνία Ζεγοβίνη. Ποιος είναι ο ρόλος που προβλέπεται εκεί για τους Βοσνίους Σέρβους. Δεύτερον, την περασμένη Σαββατοκύριακο μου στο Κάιρο. Και ανησυχώ πολύ όσον αφορά τα, τις, ε, τα επεισόδια που ήταν στο Αλάσκα αυτό είναι κάτι που έχει επιπτώσει στον ομοαμεθυνικό κόσμο και όχι μόνο στους Παλαιστινίους και δημιουργεί και προβλήματα σε μετριοπαθείς μου αμεθανούς. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. Το λόγο για ένα λεπτό στον συνάδελφο Γκόμες, στην συνάδελφο Γκόμες. Και μετά κλείνω τον πρώτο γύρο ερωτήσεων για να απαντήσει ο Υπουργός. Παρακαλώ. Uh, Καλωσορίσατε, ορίσατε κύριε Υπουργέ για τη Μέση Ανατολή. Δεν είπατε τίποτα για την Ισραηλινή γραμμή για τις εγκαταστάσεις. Ε, δεν παίζει πια ρόλο αυτό. Δεύτερον για το Αφγανιστάν. Τι γίνεται για να αναθεωρηθεί αυτή η πολιτική των ΗΠΑ που δεν την αναθεωρούν όπως σκοπεύανε. Αναφερθήκατε παραδείγματο στι επιπτώσει που θέλουμε να υπάρχουν για την κοινωνία των πολιτών. Αλλά ε, ο τομέα τη δικαιοσύνη απέσχε και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχαριστικό. Τρίτον, Στρι Λάνκα δεν τέθη το θέμα της ε, διακοπής του GSP Plus. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην Υπουργό για να μας απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω θεματικά. Δεν θα απαντήσω σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά και θα αρχίσω εκφράζοντας τη λύπη μας για την απώλεια των ζώων των Βρετανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν. Πάντοτε είναι εξαιρετικά ε, λυπηρό όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά επίσης και για τις οικογένειες τους. Αρχίζω λοιπόν με το Αφγανιστάν για να πω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 35.000 ανθρώπους εκεί. Είναι η μεγαλύτερη αποστολή. Κάποιος διακόπτει χωρίς μικρόφωνο. Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να πει η Προεδρεύουσα. Είναι μια μεγάλη παρουσία και βρισκόμαστε εκεί με μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. Και αυτό το οποίο συζητήσαμε είναι μια ευρύτερη παρουσία, όχι μόνο στρατιωτική που είναι σημαντική και θα συνεχιστεί στο προβλέψιμο μέλλον, αλλά επίσης το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους Αφγανούς να οικοδομήσουν τη χώρα τους, να ανακτήσουν μεγαλύτερη ιδιοκτησία της όλης διαδικασίας ε, αποκατάσταση της κοινωνίας των πολιτών κατά πολέμηση της διαφθοράς. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα πάρει χρόνο, αλλά πρέπει να συμβεί. Και βαθμία υποστηρίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση και ο πρόεδρος Καρζάη θα λειτουργήσουν σε ευρύτερη βάση και τώρα που επανεξελέγει ο πρόεδρος θα έχει την ισχύ να τα αντιμετωπίσει. Ε, ε, βεβαίως η προσοχή ε, εστιάζεται στην ασφάλεια αλλά επίσης και στο κράτος δικαίου και η Προεδρία καταβάλει προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής και στη διάσκεψη κορυφής συζητήθηκε και στη συνάντηση με την Αμερικανική κυβέρνηση όπου το θέμα Αφγανιστάν-Πακιστάν ήταν στην ατζέντα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δει κανεί την περιφερειακή διάσταση αυτής της σύγκλουσης. Η κατάσταση στο Πακιστάν είναι διαφορετική, αλλά επηρεάζει η, μία κατάσταση στην άλλη και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και ασφαλώς θα συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι τώρα έχουμε θέσει το πλαίσιο για μια πολύ πιο συνεκτική νέα στρατηγική που θα ενισχύσει την πολιτική διάσταση, την ε, ανάπτυξη της δημοκρατικής κοινωνίας ε, πολύ περισσότερο ε, από τη στρατιωτική διάσταση. Ναι, εχθές ε, υπογράφηκε η συμφωνία και η συμφωνία Μάλλον εχθές ο κύριος Κλάους υπέγραψε την απόφαση και τώρα από 1η ε, Δεκεμβρίου θα τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία και επίσης ήδη αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για τα δύο άτομα τα οποία θα οριστούν. Δεν θέλω να κάνω βλέψεις, Μόλις ε, ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, ο κύριος Ράμφερ, το πρόεδρος Συμβουλίου, θα ε, συγκαλέσει μια έκτακτη διάσκεψη κορυφής θα, ευρύ, θα είναι κάπου στα μέσα του Νοεμβρίου, δεν έχω ακόμα ημερομηνία. Εν πάση περιπτώσει όλα θα είναι έτοιμα για να λειτουργήσουν πρώτης δωδεκάτου. Σχετικά με τη χρηματοδότηση του κλίματος. Ε, πράγματι έχουμε μια ευρωπαϊκή εντολή και αυτό είναι πολύ καλό από πλευράς Προεδρίας ελπίζαμε ότι θα επιτύχουμε κάτι παραπάνω, περισσότερη εξειδίκευση. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει το πλαίσιο για την ανάγκη χρηματοδότησης, ουσιαστικής χρηματοδότησης. Ε, έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα αρθούν τα εμπόδια, τα εσωτερικά εμπόδια για την ανάπτυξη ε, μηχανισμών λειτουργίας, Ο καθένας θα συνεισφέρει ανάλογα με το ΑΕΠ του και ανάλογα με τις εκπομπές του και οι φτωχότερες ε, χώρες θα δεχθούν υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι χώρες του παραρτήματος 1 οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία κλπ. κλπ. πρέπει και αυτές να αναλάβουν μεγάλο μερίδιο της χρηματοδότησης εν ώψη της Κοπενχάγης. Νομίζω ότι έχουμε μια ισχυρή εντολή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ακόμα ηγέτες αυτής της όλης ε, προσπάθειας. Σχετικά με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι, η Κομισιόν συνιστά να ξεκινήσει η διαδικασία και να δοθεί μια ημερομηνία. Το ζήτημα του ονόματος δεν έχει επιληθεί, αλλά η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει εμπλακεί πολύ σοβαρά στην υπόθεση αυτή και ελπίζουμε ότι το Δεκέμβριο θα έχουμε κάποια πρόοδο επ' αυτού. Επίσης, σχετικά με το Κωσυφοπαίδιο. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν αποτελούσε μέρος των πρώτων συζητήσεων. Τώρα ε, θέλουμε Σερβία, Μαυροβούνιο και Φιρόμ να βοηθήσουν και να περιληφθούν και αυτά στη συζήτηση μαζί με την Αλβανία και την Βοσνία να βοηθήσουμε όλους να προλάβουν ώστε να μην καθυστερήσουν. Και το Κωσυφοπαίδιο βρίσκεται στο πλαίσιο των συζητήσεων, αλλά εκεί η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη λόγω της ειδικής κατάστασης που επικρατεί. Πάντως είμαστε στη διάλογο με το Κομισιόν για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτό το ζήτημα και θα υπάρξει μια έκθεση προοδού στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν μπορώ να επανέλθω από αυτού τον Δεκέμβριο. 10-11 Δεκεμβρίου. Τι άλλο λέει ο Υπουργό. Yes, I believe that, that, um, Syria saw the... Συρία. Ναι, η Συρία είδε τα οικονομικά ωφέλη της υπογραφής μιας ε, συμφωνίας δηλαδή προηγουμένως ανησυχούσε για ε, την απώλεια ε, τελών και ε, εσόδων από τα από τους φόρους και τα τέλη, ωστόσο διαπίστωσε ότι είναι προς το συμφέρον στο ελεύθερο εμπόριο. Σερβία. Υπάρχει, συνεχίζεται η συνεργασία, υπάρχει διαδικασία στο Διεθνές Δικαστήριο σε άλλους τομείς σημειώνεται πρόοδος, αυτό βοηθά. Είναι σημαντικό οι χώρες στην περιοχή να δείχνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, επιτεύγματα, ότι η προσπάθεια αποδίδει ώστε να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις υποσχέσεις της. Απαντώντας το Μεσανατολικό, όχι, δεν συζητήθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση το ζήτημα των υποδομών, των Αποχέτευση και λοιπά ε, της όλης υγιεινής τέλος πάντων δεν συζητήθηκε ωστόσο η κατάσταση είναι γνωστή στο Συμβούλιο και βρίσκεται πάντοτε επιτάπητο στο ζήτημα αυτό σε όλες τις συνεδριάσεις. Ονδούρας. Τι μπορώ να πω. Ναι, παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά. Έχει εκδώσει το, η Προεδρία δήλωση και έχουμε συζητήσει ε, πιθανές, πιθανά σενάρια αν δεν υπάρξει συμβιβαστική λύση. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν, περιμένουμε τι ακριβώς θα συμβεί στην Ονδούρα. Πάντως παρακολουθούμε στενά και πιστεύω ότι και η Ισπανική Προεδρία με τη σειρά της ε, θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά την κατάσταση. Συνεχίζουμε με το δεύτερο γύρο των τοποθετήσεων. Για ένα λεπτό κύριο Πέτερινγκ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα για άλλη μια φορά να επανέλθω στο θέμα τη Μέσης Ανατολή και στην ερώτηση τη συναδέλφου Κόμερ. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμασταν και είμαστε πάντα ένα τίμιος ε, διαμεσολαβητής όσον αφορά και το Ισραήλ αλλά και την ε, ε, αξιοπρέπεια της Παλαιστίνης. Προσπίζουμε το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να μπορεί να αναπτυχθεί αξιοπρεπές Παλαιστινιακό κράτος. Δεν αρκεί να πούμε τώρα ότι είναι γνωστή η στάση για τις επικίσεις Προφανώς αυτή τη στιγμή η Αμερικανική κυβέρνηση αλλάζει τι τάσει τη από ό,τι βλέπουμε και θα ήθελα να παρακολουθήσω την Προεδρία να πει δημόσια και ξεκάθαρα ότι δεν θα βοηθήσει στην ειρήνευση τη μέση Ανατολή το να συνεχιστούν οι εγκαταστάσει αυτές των οι επικισμοί των Ισραηλινών. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σας ένα λεπτό. Thank you. Um, ναι, σας ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση και το σχετικό έγγραφο. Λέγεται ότι υπάρχει μια κατανομή ε, εργασία για τον προγραμματισμό των γεωγραφικών ε, και άλλων ε, μέσων που θα πρέπει να οργανωθεί μέσα στα πλαίσια του 2009. Εκπλήττομαι γιατί θα πρέπει καταρχήν να έχουμε μια πρόταση από τον το εκπρόσωπο που δεν έχει ακόμα οριστεί. Πώς βλέπετε εσείς λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Και θα ήθελα επίση να επανέλθω στην ερώτηση της κυρίας Κόμους για το GSP Plus στη Σρι Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πότε θα πάρουμε ε, μια απόφαση για την διακοπή αυτής της ενίσχυσης. Τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε στο διάλογο με την Λιβύη και το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε τα πιο επίκαιρα των στοιχεία για την διαπραγματεύσεις με την ε, Συρία και τη Λιβύη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Μπράτνερ. Ο κύριο, κύριος Τάνοφ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Α, να ρωτιόμαι κύρια Πρόεδρε, κατά πόσον εξετάστηκε το θέμα της διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας που επίκειται και το ιδίως το θέμα ότι η Ρωσία ε, επιμένει να υποστηρίξει το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ότι ετοιμάζονται να πουλήσουν πυράβλους S300 στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Επίσης, ο νέος υπότος εκπρόσωπος, όποιος και όποια να είναι, θα είναι ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εγώ έχω όμως αντιφατικές απαντήσεις από διάφορους υπαλλήλου. Είναι η άποψη του ε, Συμβουλίου ότι θα πρέπει να έρχεται εδώ ενώπιόν μας και για επικύρωση, μια που θα είναι υποψήφιος και για αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Τάνο, Πρόεδρος. Συνάλφος Λέζινγκ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση για την Αφρική. Υπήρξε και ένα ψήφισμα του Συμβουλίου για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών σχετικά με το Κονγκό και στη δήλωση αυτή αναφέρεται ότι δεν είναι μόνο ομάδες επαναστατών αλλά και ε, ο κογκολικός στρατός ε, καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτός ο στρατός όμως εκπαιδεύεται από την ΟΙΖΕΚ Κόγκο. Αυτό τι σημαίνει ότι η ΟΙΖΕΚ στις προσπάθειές τους ε, για την ε, μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφαλείας έχει αποτύχει. Εσείς κυρία Υπουργέ πώς αξιολογείτε την επιτυχία της ΟΙΖΕΚ. Και μία παρόμοια ερώτηση για το Πακιστάν. Στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βοηθήσει στην δημιουργία μονάδων κατά των τρομοκρατών, αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε πολλά πράγματα. Τι προβλέπετε ακριβώς σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ρε Το λόγο για ένα λεπτό στον Αλφα Λαντσπέργκης. Δύο απλές ερωτήσεις για τη Γεωργία, Πρόεδρε. Η Προεδρέα παρακολουθεί την πρόσφατες εξελίξεις με την στάση της ε, Ρωσίας στο τομέα αυτό που είναι κάποιες ε, περιβαρισκευικές δράσεις για στρατιωτικές δράσεις μετά. Και δεύτερον, ποια είναι η στάση ε, ποιος είναι ο λόγος της τάσης των Ισπανών ε, αρχών που δεν δίνουν θεωρήσεις στα διαβατήρια γεωργιανών δικηγόρων. Η Προεδρία προτίθεται να ξεπεράσει αυτά τα τεχνικά εμπόδια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λετσπέργης. Το λόγο έχει η συνάδελφος Ρία Λίντσεν για ένα λεπτό. Mm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω να σας υποβάλω μια ερώτηση πάνω σε ένα σημείο το οποίο έχουμε ήδη αναφέρει όταν μας είχατε σας είχαμε επισκεφτεί ως εκπροσώπους του Πολωνικής ε, Βουλής. Πρόκειται για το θέμα της εταιρική σχέσης στην ανατολικές χώρες. Πώς βλέπετε εσείς την ε, προοπτική μετά από την Προεδρία σας ε, όσον αφορά τη δέσμευση των χωρών που πρόκειται να καλυφθούν από αυτό το πρόγραμμα. Ιδίως αναφέρομαι στη Λευκορωσία. Η Προεδρία πώς βλέπει τη δυνατότητα η κοινωνία των πολιτών εκεί να συμπεριλάβει και την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας δηλαδή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Εγώ μόλις επέστρεψα από την Παλαιστίνη με την αντιπροσωπεία την προηγούμενη εβδομάδα και πρέπει να σας πω ότι ο επικισμός συνεχίζεται εμείς ε, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ε, είδαμε με τα μάτια μας 53 άτομα μιας οικογένειας να απελάβνονται, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, και να εγκαθιστούν μπροστά στα μάτια μας ε, επίκους. Ε, λοιπόν, είδαμε τα μάτια μου καταστροφές σπιτιών και το τείχος να μεγαλώνει, τσιμέντο παντού. Λοιπόν, απέλαση, ε, αγροτών στην Υπεριορδανία. Τι γίνεται. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη Συμφωνία Ελευθέρων Ανταλλαγών, Ανταλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ. Λοιπόν, πώς θα αποκλείσουμε από αυτές τις συμφωνίες τα αγροτικά προϊόντα των επικισμών η συνάδελφος Μούνιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, εγώ δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά άκουσα ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα σχετικά με τη Γεωργία. Το λέω αυτό ότι πραγματικά δηλαδή δεν μπορεί να λέμε τέτοια πράγματα για την ισπανική κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν ο κύριος Λαντσμπέργης θέλει να πει κάτι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ απαράδεκτη την ορολογία που χρησιμοποίησε για την ισπανική κυβέρνηση η οποία θα σκίσει και την προεδρία εντός ολίγου. Ευχαριστώ κυρία Μουνιώθ. Η κυρία Φλότρο για ένα λεπτό. Καλημέρα κυρία Μέλστρομ, μεγάλη χαρά να σας ξαναβλέπουμε εδώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, Συρία. Μου φάνηκε να κατάλαβα ότι η Συρία υπέγραψε τη Συμφωνία Συνεργασίας, που δεν το ξέρα μέχρι τώρα, Τώρα μιλάτε εσείς ε, για ελεύθερες ανταλλαγές ε, που ε, έδωσαν νέα απνοή στην υπογραφή της συμφωνίας με τη Συρία κτλ. Αλλά ξέρετε τα προβλήματα των βουλευτών δεν ήταν το θέμα των ελευθέρων ανταλλαγών, ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πού βρίσκονται λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη συμφωνία, στην υπογραφή, τέλο πάντων τη συμφωνία συνεργασία υπάρχει μία απέτηση που θα λέει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη Συρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεύτερον θα έχουμε και εκλογέ στην Τινησία. Εντό εισαγωγικών το λέω οι εκλογές βία, εξαφανίσεις, ε, ε, οχλήσεις, ε, φυλακίσεις των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το φρικτό, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Λοιπόν, η Προεδρία μπορεί να αντιδράσει επί τόπου μέσα από τις αντιπροσωπείες που έχουμε εκεί, ας πούμε την αντιπροσωπεία της Κομισιόν. Μπορούμε τέλος πάντων να πούμε ποιες είναι, ότι το απαιτούμε δηλαδή να σταματήσει αυτή η απέσια κατάσταση η οποία συνεχώς υποβαθμίζεται μπροστά στα μάτια μας. Νόιζερ για ένα λεπτό ολοκληρώνει το δεύτερο κύκλο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ ξανά σε κάτι που θύθεξε. Είχαμε ρωτήσει πώς αξιολογείτε εσείς τη γνωμοδότηση του νέου Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας ότι στο Αφγανιστάν έχουμε μια κατάσταση εμπόλεμη. Συντυχώς δεν μας απαντήσετε σε αυτό. Και δεύτερον, απόρρισα που είπατε ότι ο πρόεδρος Καρζάη επανεξελέγει. Μα εμείς είδαμε όλοι ότι ο πρώτος γύρος ε, ήταν αντικείμενο νοθείας και ο δεύτερος γύρος δεν έγινε. Πώς εξελέγει τότε. Ευχαριστώ κύριε Νόιζερ. Θα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει. Yes, thank you. I can see that the... Ευχαριστώ. Η ποικιλία των ερωτήσεων δεν άλλαξε από τότε που ήμουν εγώ εδώ μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζω κύριε Πότερινγκ και απαντάω και σε άλλους, γνωρίζω τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αφοσίωση στο θέμα ε, της Παλαιστίνης, της... και επίσης και τη δική σας προσωπικ... το δικό σας προσωπικό ενδιαφέρον και δέσμευση. Ναι, Υπουργό Εξωτερικών έκανε ένα βήμα πίσω λέγοντας ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει στο Ισραήλ. Στο θέμα της Ιερουσαλήμ, η Προεδρία έκανε μια δήλωση και παραθέτω. Η Προεδρία ε, ε, επιμένει ότι η ε, οι καταστροφές των ε, σπιτιών, οι μετακινήσεις ε, δεν συμβάλλουν στην επίλυση της ε, σύγκρουσης του ζητήματος και επίσης δηλώσαμε ότι είπαμε ότι τα προϊόντα από τους επικισμούς που προέρχονται από τις περιοχές των επίκων δεν μπορούν να είναι να περνάνε ελεύθερα από το Τελωνείο. Ε, επιμένουμε στη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ και λέμε ότι το Ισραήλ είναι η 67η ε, ε, ε, το Ισραήλ βρίσκεται στα όρια που ήταν και το 1967 και φυσικά δεν συζητούνται θέματα τα οποία προέρχονται από τα κατευχόμενα. Για τη Σριλάνκα τώρα. Το, οι αρχές της Σριλάνκα δεν έχουν εφαρμόσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Άρα λοιπόν ο διάλογος μαζί τους πρέπει να συνεργαστεί και τώρα το θέμα συζητείται στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και παρακολουθούμε το θέμα από κοντά. Ρωσία. Δεν συζητήθηκε το, η Ρωσία γενικότερα. Στην ε, mini ε, session θα, συζητηθεί, θα συζητηθούν τα θέματα σχετικά με τη Ρωσία και βεβαίως και στην διάσκεψη κορυφής με την Ρωσία και μετά βεβαίως θα υπάρξει και αναφορά στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι αρχές περιλαμβανομένες και της εδαφικής ακαιρεότητας της ε, Γεωργίας και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να πιστεί η Ρωσία ότι δεν είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον στη φάση αυτή να στρατιωτικοποιείται το Ιράν με δική της βοήθεια. Ωστόσο, τα γενικότερα ζητήματα με τη Ρωσία θα συζητηθούν σε απότερη φάση. Λεύκο Ρωσία. Από πλευράς Σουηδικής Προεδρίας ε, είχαμε μια συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών, με εκπροσώπους, των, με εκπροσώπους ε, πολιτών της αντιπολίτευσης και επίσης όταν δρομολογήθηκε η εταιρική σύμπραξη προς Ανατολάς ε, ε, κάναμε μια σημαντική προσπάθεια μαζί τους όπως συμφωνήσαμε και με τον κύριο Λίζεκ να δούμε αναζητούμε τρόπους ώστε να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία των πολιτών στην Λευκορωσία. Και βεβαίως η Λευκορωσία θα βρίσκεται πάντα στην ατζέντα του Συμβουλίου. Ο ύπατος εκπρόσωπος βεβαίως είναι ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν λοιπόν διοριστεί θα έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ακρόαση όπως ακριβώς και όλοι οι υπόλοιποι. Και επίσης στη συνθήκη αναφέρεται ότι οι απαραίτητες επαφές θα πρέπει να γίνουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως θα εξαρτηθεί από το πότε θα οριστεί το άτομο αυτό και πότε είναι δυνατό το άτομο αυτό να έρθει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε σε επαφή με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και με τον κύριο Μπούζεκ για να δούμε πώς θα επικοινωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη στιγμή που θα καταστεί σαφές ποιο θα είναι το άτομο αυτό, ποιο ή ποια. Και θα έρθει βεβαίω αυτός ή αυτή στο κοινοβούλιο. Και επίσης θα θεσπίσει και το πλαίσιο, πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Ποιο θα είναι η ε, στελέχωση, το πεδίο δράσης, ε, ε, όλα αυτά θα πρέπει να καθοριστούν. Δηλαδή όταν οριστεί ο ύπατος εκπρόσωπος και όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και μετά από σε βάθος συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά θα οριστικοποιηθούν όχι αργότερα από τις 10 Απριλίου 2010. Τι άλλο. Νομίζω ότι ο πρόεδρος άρχισε την ομιλία του επισημένοντας ότι η Συρία υπέγραψε και εγώ θυμάμαι τις συζητήσεις σε αυτή την Επιτροπή και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Συρία. Πάντοτε υπήρχαν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη Συρία και ε, υπήρχε πάντοτε θέμα συζήτησης από αυτού μαζί τους. Και έγινε και μια ξεχωριστή δήλωση που υπογραμμίζει τη σημασία που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. αυτό έρχεται ως προστίκη, δεν ε, τροποποιεί τη συμφωνία, αλλά έρχεται ως προστίκη και ως ε, υπογράμμιση, ας πούμε, της συμφωνίας. Σχετικά με το Κονγκό, ίσως δεν κατάλαβα καλά Ε, πρέπει να το ξαναδώ γιατί δεν μπορώ να σας δώσω σήμερα απάντηση από αυτού. Νομίζω αυτά κύριε Πρόεδρε. Α, για τη Γεωργία δεν είπατε λέει κάποιος από το ακροατήριο. Ήταν το θέμα της εδαφικής ακερότητας της Γεωργίας μου ρωτήσατε. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Προεδρεύουσα. Αναφερόμουν, αναφερόμουν σε πρακτικές εκφοβισμού που και προπαγανδιστικές προσπάθειες σχετικά με τη χορήγηση θεώρησης διαβατηρίων που μπλοκάρονται από την Ισπανία. Δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο άλλοι άνθρωποι που έχουν παράνομα ρώσικα διαβατήρια μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ οι Γεωργιανοί με νόμιμα διαβατήρια δεν το πράττουν. The, the of, of... Ναι, βεβαίω. Τονίσαμε την ε, αρχή της εδαφικής ακαιρεότητας, αυτό προς την Ρωσία και σχετικά με την ε, σύνδεση και το θέμα χορήγησης ε, θεωρήσεων βρίσκεται επί Ίσως ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς ελέγχθη στη Μαδρίτη και δεν έχω μπροστά μου την απόφαση. Ωστόσο, ε, πράγματι το ζήτημα αυτό εκκρεμεί και θα συζητηθεί και πάλι το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όταν θα κάνουμε και μια γενικότερη αξιολόγηση τη ανατολική εταιρική σχέση. Θα ήθελα να τονίσω ότι και στην δική μου ερώτηση για το Πακιστάν δεν δώσατε καμία απάντηση. Δεν απαντήσετε σε καμία από τι δικέ μου ερωτήσει. Θέλω να το σημειώσετε. Eh. Τέλειωσε η συζήτηση. Και αυτή η πτυχή δεν έχει προβλεφθεί, ε, δεν έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστούμε λοιπόν την Υπουργό για όσα μας είπε. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο, να εμβαθύνουμε σε επόμενες συνεδριάσεις ε, όσα δεν μπορέσαμε να εμβαθύνουμε σήμερα στο επανειδήν. Συνάδελφοι σας παρακαλώ. Να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο. Λοιπόν, αν κάποιος από τους παρόντες θέλει να φύγει από την αίθουσα, να το κάνει σύντομα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, σε ένα κλίμα ήρεμο και όχι ταραγμένο από τις οχλήσεις της εθούσης. Λοιπόν, έχουμε την έκθεση για την τροποποίηση του μηχανισμού σταθερότητας. Η κυρία Μπράντνερ έχει το λόγο, η Φραντσίσκα Μπράντνερ έχει το λόγο. Um, yes, thank you. I think it's a bit... Uh, Σας ευχαριστώ. Κάπως έχει πολύ φασαρία, Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν ενδιαφέρονται για τις εργασίες μας και βρίσκονται στα πρόθυρα της εθούσης καλά θα κάνουν να φύγουν για να μπορέσουν να εργαστούμε με την ησυχία μας. Εάν θέλετε να μείνετε εδώ και να δουλέψετε, καθίστε ήσυχα, αλλιώς συνεχίστε τη φλιαρία έξω. So we are speaking today about the stability instrument. Αναφερόμαστε στο μηχανισμό σταθερότητας που είναι ένα δημοσιονομικό μέρος για την αντιμετώπιση των κρίσεων και για την δίνευση. Και θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία και να το εξηγήσω και μετά να εξηγήσω και στους που έχουμε εισαγάγει μέχρι στιγμή και να δώσω μια γενική εικόνα γιατί συζητάμε. Είναι δύσκολο, πρόεδρο, όταν κάνει τόσο φασαρία στην αίθουσα. Τις πάντων. Αυτό το μέσο σταθερότητας λέγεται ξεκάθαρα στην νομοθεσία ότι είναι συμπληρωματικό σε μέτρα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόθεση κοινή ε, εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφαλεία και του στόχου τη. Είναι συμπληρωματικό λοιπόν, δεν είναι τμήμα τη ε, ΚΕΠΑ. Έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούνται ε, σχέδια σε δύο κυρίω καταστάσει. Η μία είναι κατάσταση κρίσης και ενάρξης κρίσης, δηλαδή οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα του να περάσουν διαμάχη και προβλέπεται ότι θα υπάρχει κρίση σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν, δεν προγραμματίζεται τον των προτέρων, αλλά βέβαια μπορεί κανένας να μαντέψει που θα υπάρξει προσεχώς μια κρίση και αυτό είναι το πιο μεγάλο τμήμα του προπολογισμού. 73% δηλαδή για τις καταστάσεις αυτές κρίσης και ενερχόμενες, ε, ενερχόμενων κρίσεων. Η Κομισιόν και τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για την αντιμετώπιση και άλλων κρίσεων. Το πρώτο. Το δεύτερο που έχουμε, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, είναι όχι κρίση, σταθερή κατάσταση, αλλά για την ανεπτώση συγκεκριμένων ε, παγκοσμίων και διαμεθοριακών ε, εντάσεων. 27% του προπολογισμού προβλέπεται εδώ. Και αυτό το τμήμα καλύπτεται από το άρθρο 4 και έχει τρεις κυρίους ε, τομείς παρέμβασης. Ο πρώτος είναι η απειλή στο κράτος ε, δικαίου, στην δημόσια υγεία και στη δημόσια υποδομή. 7% προβλέπεται εδώ. Και η δυνατότητα παρέμβασης εδώ είναι πολύ ευρεία, δηλαδή αντιτομοκρατία, δημόσια υγεία και πολλά άλλα. Και μετά υπάρχει και μια δεύτερη γραμμή κάτω από το τμήμα αυτό των σταθερών όρων, δηλαδή χημική, ραδιολογική και πυρηνική απειλή. 15%. Και το τρίτο είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων πριν και μετά την κρίση. Και αυτό αφορά μακροπρόθεσμα μέτρα, ανάπτυξη της λογόμενης η Ειρηνή μέσω της εταιρική σχέσης που θα ακούσατε ίσως κάπου. Είναι μια εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών που δεν αναφέρεται στο αρχικό κείμενο, αλλά έχει καθοριστεί με μια επιστολή της ε, Εκτελεστικής Επιτροπής. Ε. Έγινε μια αναθεώρηση, μια νέα στρατηγική, αλλά αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνεργασίας της Κομισιόν με την κοινωνία των πολιτών. Μακροπρόθεσμα. Οι τροπολογίες που έχουμε προετοιμάσει μέχρι στιγμής, η πρώτη ας πούμε, είναι να αναγνωρίσουν ε, ειρηνικά ε, ρητά αυτή την ελληνική ε, εταιρική σχέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μια πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Και θέλουμε την αναγνώριση αυτή να αναφέρεται στο νομοθετικό κείμενο. Η δεύτερη τροπολογία αφορά τις προτάσεις Κομισιόν. Η Κομισιόν προτείνει αύξηση της χρηματοδότησης σε σταθερές, σταθερούς όρους, όπως σας είπα, από 7% στο 10%. Να χρησιμοποιούν δηλαδή περισσότερα χρήματα στον τομέα αυτό. Σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι οι προτεραιότητε που θέλει να ορίσει η Κομισιόν. Γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει τα περαιτέρω αυτά χρήματα, γιατί το μέσο είναι πάρα πολύ ευρύ και θέλω κάποιε ενδείξει εκ των προτέρων πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Ιδίω για το τι το ειδικό άρθρο είναι πάρα πολύ ευρύ. Οι άλλε τροπολογίε αφορούν το τελευταίο τμήμα, το 4-1 δηλαδή, Και θα σας διαβάσω, λέω, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών και τη συμμετοχή της στην πολιτική διαδικασία συμπεριλαμβανών μέτρων για να ενδυναμώσουν τον ρόλο των γυναικών και να προωθηθεί ανεξαρτησία, πλουραλισμός και επαγγελματισμό των μέσων ενημέρωσης. Και θα σας πω γιατί το έχουμε προσθέσει αυτό. Γιατί υπάρχουν κάποια χρήματα για την υποστήριξη των γυναικών και των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης μέχρι να φτάσουμε σε μια ειρηνική συμφωνία. Αλλά μετά δεν προβλέπεται τίποτα. Και πρέπει να δώσουμε τα χρήματα για να προωθήσουμε τον ρόλο των γυναικών. Στη μεταβατική φάση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τίποτα. στην φύση κατά καθορίζεται το Σύνταγμα, καθορίζει διάφοροι οργανισμοί που υπάρχουν. Υπάρχει κίνδυνο οι γυναίκε να χάσουν. Και επίση θέλουμε και επαγγελματικά μέσα ενημέρωση για να προωθηθεί αυτή η διαδικασία εκδημοκρατισμού. Σε αυτή τη μεταβατική φάση νομίζω θα πρέπει να υποστηριχθούν αυτά τα δύο ε, σημεία. Και εκεί θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο το μέσα αυτό σταθερότητα. Αυτέ είναι οι τροπολογίε μέχρι στιγμή και θα ήθελα επίση να τονίσω μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν και που αφορά το θέμα των μικρών όπλων και ελαφρών όπλων. Αυτό είναι κάπως μια διαμάχη μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγχει η ΚΕΠΑ, η κοινότητα, μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φτάσανε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι η Κομισιόν επιτρέπεται να εργάζεται για τα μικρά και ελαφρά αυτά όπλα. Το θέμα που ήθελα τώρα είναι πού είναι η κατανομή ε, εργασίας μεταξύ Εκτελεστικής Επιτροπής και Συμβουλίου. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια πολιτική δήλωση, κοινή εργασία, συνένεση δηλαδή, πώς συνεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό αντί να καθόμαστε να τσακωνόμαστε για μικρά άκαμπτα κείμενα. Θα ήθελα λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο θα εξακολουθεί να εργάζεται στο τομέα αυτό και όχι μόνο η Κομισιόν που έχει τώρα πίσω τη συναπόφαση του δικαστηρίου και θέλουμε να βρούμε έναν καλό τρόπο για να λύσουμε τα προβλήματα και τώρα που θα υπάρχει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα είναι γελίο να κατασπαταλάμε βδομάδες για το θέμα αυτό προκαταρτικά. Και ήμουνα σε επαφή με την Εκτελεστική Επιτροπή και το Συμβούλιο ανεπίσημα για τα θέματα αυτά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε με τρόπο που να μπορέσουμε να μην αυξηθεί η σύγκρουση μεταξύ των ε, κοινοτικών οργάνων, πράγμα που μειώνει η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ε, ε, ευχαριστώ την κυρία Μπράντνερ. Αρχίζει η συζήτηση. Η κυρία Λέζινγκ, συντονίστρια της Γκου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι βέβαια πολλοί τομεί ε, του μέσου αυτού είναι πολύ θετικοί και τους ε, θεωρούμε πολύ θετικούς παραδείγματος χάρη η ενίσχυση που δίνεται για τα παιδιά στρατιώτες. Πολλά πολύ θετικά πράγματα υπάρχουν. Έχουμε όμως κάποια ουσιαστικά προβλήματα εδώ γενικού τύπου αρχής. Το ένα είναι πώς ορίζουμε την κρίση εδώ. Κατά τη γνώμη μας, αυτός ο ορισμός της κρίσης είναι πολύ ευρύς. Δεν ξέρω, επίτηδες έχει γίνει αυτό, εσκεμένα, ότι σχεδόν κάθε, κάθε κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ως κρίση. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εμείς στην ΚΟΕ είναι ότι ε, αναμειγνύονται εδώ η κοινωνία των πολιτών με θέματα της ε, ε πολιτικής άμυνας. Ξέρουμε ότι γίνεται, θέλουμε να το επικρίνουμε. Επίσης θέλουμε να επικρίνουμε τον προστατορισμό του μέσω αυτού στα ίδια οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω εδώ και κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Θα σας τη διαβάσω γιατί συμπεριλαμβάνει κάποιους αριθμούς. Η συνάδελφος Μπράτνερ τόνισε ότι η τροπολογία προβλέπει τα, με, τους πόρους για τα μέτρα αυτά βάσει του α, άρθρου 4.1 του κανονισμού να αυξηθούν από 7 στα 10%. Στο άρθρο αυτό ε, συμπεριλάβεται και η προστασία κρισίμων υποδομών, παραδείγματο χάρη ενέργεια και εμπορικών οδών, που μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται μέσα στα πλαίσια του ετησια εκθεσης έκθεσης 2009-2011. Τα προτινόμενα συμπραγματικά κονδύλια αναφέρονται στις ειδικέ ανάγκες που έχει αυτός ο τομέας και μετά για τη συνεργασία με την ΚΕΠΑ. Έχω να σας πω ότι η εμπλοκή ε, των διαφόρων τομέων είναι θετική, αλλά πώς μπορούμε να διακρίνουμε πολιτικούς στόχους από στρατιωτικούς. Μήπως είναι προβληματικό να τους αναμειγνύουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μουνίθ συντονίστρια των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ την συνάδελφο Μπρέπνερ ε, για την ε, δουλειά της και την ευχαριστώ επίσης για την ε, συνεργασία με τους σκεώδεις εισηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Είχαμε συνεδριάσεις ιδιαίτερα ειλικρινείς και αποτελεσματικές. Συμφωνεί λοιπόν η σοσιαλιστική ομάδα με τη γραμμή της εισηγήτριας και για τις δύο πρώτες ε, τροπολογίες σχετικά με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τον ε, συνεχώς ευξανόμενο ρόλο των γυναικών και στο δύο η αναφορά της ε, για την Peace Building Partnership συμφωνούμε. Συμφωνούμε διότι υπήρχε αυτό το κενό ε, στον προηγούμενο κανονισμό για το μηχανισμό σταθερότητας. Επίσης θέλουμε να συμφωνήσουμε με την Κομισιόν για να ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια διότι θεωρούμε ότι αυτό το μέσο είναι σύμβατο με, το, με όσα εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια. Ζητάμε όμως από την Κομισιόν να έχουμε ένα αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο, στρατηγικό σχεδιασμό για το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Και έχει λόγο λοιπόν, ε, έχει δίκιο συγγνώμη η κυρία Μπραντνερ να συνδέει το 3% και το υπόλοιπο 7% μέχρι να φτάσει στο 10% με αυτή την παρουσίαση των σχεδίων. Τώρα, για τις τροπολογίες της κυρίας Λόζινγκ. Δεν μπορούμε κάθε φορά εμείς να γυρνάμε στις ρίζες των πραγμάτων. Πρόκειται για κάτι το οποίο έχει συζητηθεί επί μακρόν πριν από δύο χρόνια. Λοιπόν, άμα πρέπει να ξαναρχίσουμε να ορίζουμε από την αρχή τι εστί κρίσεις, ε, ε, με, με, μετακρίσεις ή οτιδήποτε άλλο, χάσαμε την ώρα μας. Εμείς πιστεύουμε ότι θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων επί της κοινωνίας των πολιτών για τις παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε εμείς αυτά τα δύο να τα έχουμε χωριστά. Γι' αυτό δεν θα συμφωνήσουμε με την τροπολογία 5 της κυρίας Λούζινγκ. Τώρα για την 4 που αναφέρεται στα δικαιώματα του πληθυσμού, ο οποίος είναι δικιούχος του μηχανισμού σταθερότητας, μα νομίζω ότι είναι κάτι το εντελώς άχρηστο. Αυτό είναι αυτονόητο δηλαδή. Και συγχαίρω την κυρία Μπράνερ και την υποστηρίζει σοσιαλιστική ομάδα στις τροπολογίες της. Ευχαριστώ κυρία Μουνίφ η κυρία Γκόμες. Uh, η συνάδελφο Μουνή ήταν πολύ σαφή για την υποστήριξη των σημείων που έθεξε η μα. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των τροπολογιών όπου αναφέρεται στην ε, προσοχή που θα πρέπει να επιδοθεί στο ρόλο των γυναικών και θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό που είπε η συγχύτρια για την ανάγκη οι Κομισιόν και το Συμβούλιο να σταματήσουν να ε, διαμάχονται όσον αφορά ποιος είναι αρμόδος για τα θέματα των ελευθερών μικρών όπλων. Και τέλος, όπως είπε και η Μαρία Μουνής, έχω να πω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις ε, τροπολογίες της κυρίας Λούζινγκ και δεν θέλω ιδιαίτερα να σας πω ότι διαφωνώ πλήρως για την απόρριψη του συνδυασμού ε, πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων στη συνεργασία. Ακριβώς αυτή είναι μία μη ευρωπαϊκή προσέγγιση, γιατί η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι να συνδυάσουμε τα μεν με τα δε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εκπολιτήσουμε, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο το στρατιωτικό τμήμα για να μπορέσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τους σωστούς πολιτικούς στόχους και να το επιβεβαιώσει αυτό και η στρατιωτική πτυχή. Λοιπόν, δεν συμφωνούμε με αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ κύριε Αγγουράκη, εσείς είστε αναπληρωματικό μέλος ε, και έχω δυσκολίες για το χρόνο. Διότι έχω να δώσω το λόγο και σε δύο εκπροσώπους της Κομισιόν. Σας παρακαλώ δηλαδή αν μπορείτε να αποσύρετε την τοποθέτησή σας ε, ή να τα πείτε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα γιατί τελειώς δεν έχουμε χρόνο. Σε 30 δευτερόλεπτα μπορείτε να τα πείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε 5 δευτερόλεπτα θα το πω. Ε, νομίζω ότι η κυρία Λιόζινγκ έχει δίκιο όταν λέει για το θέμα των κρίσεων. Το πρόβλημα δεν είναι κατά τη γνώμη ότι γυρίζουμε πίσω. Δυστυχώς επεκτείνεται ο όρος των κρίσεων. Έχουμε αρκετές επεμβάσεις. Ήδη δεν χρειαζόμαστε ακόμα ένα σώμα για επεμβάσεις στο ιστορικό άλλων χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν, ο Δόκτωρ Καρνκούτρι και μετά ο Δόκτωρ Βόλερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες διευκρινήσεις και κάποια σχόλια από την Κομισιόν. Θα αρχίσω από τις τροπολογίες που κατέθεσε η Στι στις δικές μας τροπολογίες σχετικά με την διατύπωση για το ρόλο των γυναικών στην μετα στην ειρηνευτική διαδικασία μετά τη σύγκρουση και τις εταιρικές σχέσεις που υιοθετείται. Νομίζω ότι η συγγήτρια συμφωνεί αν πω ότι τα θέματα αυτά τα παρακολουθούμε και εφαρμόζονται από την Κομισιόν στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Ε, δεν χρειάζεται λοιπόν να περιληφθούν στον κανονισμό. Ουσιαστικά πρόκειται για πολιτική δήλωση, ώστε να υπογραμμιστεί ότι η σύμπραξη για την οικοδόμηση της ε, ειρήνης ε, θα έχει την απόλυτη υποστήριξη με χρηματοδότηση και θα περιληφθεί και στο πρόγραμμα δράσης του 2010 και αυτό θα γίνει στους προσεχείς μήνες εν ευθέτω χρόνο. Ε, και θα δείτε και το έγγραφο και θα δείτε ότι αυτοί οι τομείς καλύπτονται και επίσης ότι το θέμα της οικοδόμησης της ειρήνης καλύπτεται από το μηχανισμό. Ως προς τις ε, γυναίκες υπάρχουν ειδικά προγράμματα και κονδύλια στο άρθρο 3 με ειδικέ δράσεις ε, για τη, με βάση το ε, ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 13 και 25 και επίσης ε, με βάση το, άρθρο 4, το ψήφισμα 434 για την οικοδόμηση της ειρήνης. Αυτά είναι ούτως ή άλλως δεδομένα. Δύο πολύ σύντομα σχόλια για τις τροπολογίες και τα σχόλια που ανέφερε η κυρία Λόζινγκ. Ο ορισμός της κρίσης στο άρθρο 3.1 δεν είναι κάτι το οποίο εμείς συντάξαμε τότε. Πρόκειται για έναν τεχνικό ορισμό που βρίσκει κανείς το 1-2-1 στους ε, ε, κανόνες εφαρμογής στο, και στον κανονισμό 168. Δηλαδή αυτό ε, διευκολύνει την Κομισιόν να διαθέσει κονδύλια σε περιόδους κρίσεως για να μην ε, χρειαστεί να καταφύγει σε διεθνείς προκηρύξεις και διαγωνισμούς κλπ. τα οποία είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Και αυτός είναι ορισμός ευρύς ακριβώς για να καλύψει διάφορες πιθανότητες και σενάρια κρίσεων. Το κείμενο ήδη υπάρχει, βρίσκεται στον χρηματοδοτικό ε, κανονισμό και μπορείτε να ανατρέξετε. Μας δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε το ταχύτερο δυνατό μόλις κληθούμε. Ένα τελευταίο σχόλιο για την πολιτική και στρατιωτική πλευρά της διαχείρισης κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μέσο, για ένα μηχανισμό, για πολιτικά μέτρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν έχουμε δαπάνες στρατιωτικού χαρακτήρα. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Αυτό που κάναμε είναι το εξής. Όταν υπάρχει μια στρατιωτική αποστολή και αυτό είναι το ελάχιστο. συνήθω. έχουμε πολιτικές αποστολές, ε, αστυνομικούς, ε, ε, δικηγόρους κλπ. Παραδείγματο χάρη το 2008 είχαμε στο Τσάτ μια αποστολή στρατιωτική για να προστατευθούν οι τα στρατόπεδα προσφύγων στο Ανατολικό Τσάτ για να τους προστατεύσουμε από περαιτέρω επιθέσεις παρανόμων που έρχονταν από το Σουδάν. Και τούτο κατέστη εφικτό αρχικά μόνο με Ευρωπαίους στρατιώτες. Για, για να προσαρμόσουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα ε, με τις προσπάθειες του ΟΗΕ ε, που είχε στείλει αστυνομικούς για προστασία αυτών των ε, προσφύγων τέλο πάντων. Τότε λοιπόν αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας ε, χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό μάλιστα ε, με τις προσπάθειες του ΟΗΑ και αυτό είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου λέμε ότι λειτουργούμε συμπληρωματικά ε, σε αποστολές στρατιωτικής και πολιτικής φύσεως. Εμείς παραδείγματος χάρη εκεί ε, διαθέσαμε 30 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε τη σταθερότητα εντός της Γεωργίας, να βοηθήσουμε τους εσωτερικά εκτοπισμένους ε, πολίτες. Ο συνάδελφος ε, Βόλετ θα σας πει δύο λόγια σχετικά με το άρθρο 4 και την περαιτέρω χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο πριν περάσουμε στο 10%. Εκτιμούμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα των μικρών όπλων και ελαφρών οπλισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως Ένωση μπορεί και εφαρμόζει αυτές τις δράσεις και υπάρχει και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όταν η εστίαση είναι την πτυχή, όταν εστιάζουμε στην ανάπτυξη, τότε πρέπει να υπάρχει δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ακριβώς ιδιαίτερως εκτιμούμε την υποστήριξή σας. Τώρα, σχετικά με το αίτημα αύξηση της χρηματοδότησης ε, ε, του άρθρου 4.1 για αντιμετώπιση απειλών διεθνικών. Κάποιες τέτοιες περιοχές μπορούν να οριστούν αμέσως. Υπάρχουν δύο τομείς, δύο περιοχές όπου ε, σημειώθηκε μείωση χρηματοδότησης εξαιτίας εξαιτίας ε, μη ύπαρξης γραμμών του υποροπηρισμού. Uh, Μία γραμμή αφορούσε ε, τα ναρκωτικά και ιδιαίτερως την καταπολέμηση των οδών μεταφοράς ε, ναρκωτικών. Ωστόσο η αντιμετώπιση του ζητήματος των ναρκωτικών ε, με έναν ολοκληρωμένο τρόπο είναι μέλημά μας. Πρέπει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή γενικότερη στρατηγική. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η κατάργηση μιας άλλης γραμμής μια άλλη γραμμή άλλης γραμμής που αφορά τις νάρκες. Εδώ λοιπόν ιδιαίτερος διαπιστώσαμε ότι κάποιες δομές όπως ας πούμε σε υποστήριξη της σύμβασης της ΟΤΑΒΑ δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα μέσα. Και εδώ πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός σταθερότητας μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Ε, σχετικά τώρα με τη χρηματοδότηση με βάση το άρθρο 4.1. Το θέμα αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από του χρόνου, έχει την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αποστολή αυτού του μέσου σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. Έχουμε συζητήσει το ζήτημα των μικρών όπλων και ελαφρών οπλισμών και χρειαζόμαστε τα διαθέσιμα κονδύλια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύουμε ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου δικαιολογείται. Και μιλούμε για ένα ποσό 40-60 εκατομμυρίων. Και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Κυρία Μπράτνερ, τελειώσαμε με το χρόνο μας. Λοιπόν, πριν ψηφίσουμε στις 10 Νοεμβρίου θα έχετε όλη την ώρα για να απαντήσετε σε όλους. Αλλά λίγα δευτερόλεπτα όμως, γιατί έχουμε και το φιλοξενούμενό μας εδώ που περιμένει. 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστώ του πιο ηγητέ για το της συνεργασία και την Κομισιόν επίση για τι πληροφορίε που μα έδωσε, γιατί μου φαίνεται ότι πάρα πολύ χρήσιμη για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε όσον αφορά την συνεργασία πολιτική και στρατηγική πλευρά, νομίζω η απάντηση εδώ θαυμάσια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την ε, εμπλοκή τη και το θέμα τη ε, εταιρική σχέση. Ναι, θα πρέπει να το γνωρίσουμε. Όσον αφορά το θέμα των γυναικών, θα δούμε. Περιμένω να δω τον νέο επίτροπο για να είμαι πιο σίγουρη. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο. Ήσασταν καταπληκτικοί στη σύνθεση που κάνατε. Έχουμε εδώ τώρα τον φιλοξενούμενό μας που είναι ο αρχηγός της ε, διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Κροατίας ε, για την ένταξη. Τον καλωσορίζουμε και η έλευσή του εδώ στην Επιτροπή μας ε, συνδέεται με πολύ καλά και αισιόδοξα νέα και μάλιστα βρίσκεται εδώ διότι έπρεπε να έρθει ο Υπουργό, ο οποίο όμως βρίσκεται στην Στοκχόλμη για να υπογράψει την ε, συμφωνία με τη Σλοβενία ε, που εμπόδιζε μέχρι τώρα δηλαδή αυτή η διαφωνία με τη Σλοβενία την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας ακούσουμε λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας και να απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να ανταλλάσσω απόψεις σχετικά με τις θέσεις της Κροατίας μαζί σας. Εφτισε εξ αρχή θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμού του Υπουργού Γκόρνταν Γιάντρο Μία άλλη πολύ σημαντική ευρωπαϊκή εκδήλωση τον εμποδίζει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες ε, σήμερα. Δηλαδή συμμετέχει στην τελετή υπογραφής της συμφωνιας διετησιας Διατησίας μεταξύ Κροατίας-Σλοβενίας ε, που έγινε πριν από λίγες ώρες στην Στοχόλμη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν ε, πρόεδρε Αλμπερτίνη που μου προσφέρει την ευκαιρία να συμμετάσχω στην συνεδρίαση αυτή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι στην ατζέντα σας ε, περιλαμβάνεται, περιλαμβάνονται δύο σημαντικά θέματα, δηλαδή η έκθεση πρόοδου ε, της Κροατίας το 2009 και η στρατηγική διεύρυνση του 2009. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Κροατίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, συνεχή και πολύτιμη υποστήριξη προς την Κροατία και τον, στην πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον, την, τον εισηγητή για την Κροατία, κύριο Χάνες Βόμποντα, για την ακούραστη ε, προσπάθειά του, την αντικειμενικότητα και τις καλές συμβουλές του προς την ε, Κροατία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα προς την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψατε μου να σας παρουσιάσω τις τελευταίες εξελίξεις στην Κροατία με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων όπως επίσης και την συμμόρφωση προς τα κριτήρια ένταξης. Το περασμένο μήνα γιορτάσαμε την τέταρτη επέτειο της έναρξης, της επίσημης έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κροατίας. Θα ήταν ένα συμβολικό γεγονός, ωστόσο χαρακτηρίζεται από δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, την παραμονή της επαιτίου και μετά από σημαντική καθυστέρηση η Κροατία άνοιξε ή ε, προσωρινά έκλεισε 11 κεφάλαια συνολικά στην ε, διακυβερνητική διάσκεψη. Αυτή λοιπόν η διακυβερνητική υπήρξε η πιο σημαντική μέχρι στιγμής. Και τούτο κατέστη δυνατό όχι μόνο εξαιτία της τεράστιας, της ε, μεγάλης προσπάθειας και της δουλειάς που καταβάλαμε σε σχέση με τα κεφάλαια αυτά, αλλά επίσης επειδή υπήρξε αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Πρωθυπουργών Κροατίας και Σλοβενίας ε, βάσει ενός ανανεωμένου διαλόγου μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας και σε πνεύμα καλής γειτονίας και αμοιβαίου σεβασμού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Κροατίας προς τις Προεδρίες της Γαλλίας, Τσεχίας, Σουηδίας και τον Επίτροπο Ρεν, όπως επίσης και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειες που καταβάλουν και υποστηρίζουν και υποστήριξαν τη την επίλυση του ζητήματος αυτού και την πρόθεση της ενταξιακής μας διαδικασίας. Σήμερα στη Στοκχόλμη οι πρωθυπουργοί μας ε, υπέγραψαν μια συμφωνία διατησίας, παρουσία του Σουηδού Πρωθυπουργού. Τούτο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την αναζήτηση λύσης που θα είναι ένα κέρδος για όλους, για την Κροατία, τη Σλοβενία και για την Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει, ωστόσο ε, είμαστε αισιόδοξοι. Αξιότιμα μέλη, η Κροατία έλαβε την πιο θετική έκθεση προόδου μέχρι στιγμής και είμαστε ικανοποιημένοι που η Κομισιόν αναγνωρίζει σαφώς τα επιτεύγματά μας. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι οι ενταξιδικές διαπραγματεύσεις της Κροατίας μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στο 2010. Μας ενθαρρύνει ιδιαιτέρως αυτό, διότι η Κομισιόν προτείνει και ένα πακέτο χρηματοδότησης. Επίσης, χαιρετίζουμε τη σύσταση της Κομισιόν για συγκρότηση μιας ad hoc τεχνικής, ε, μιας ad hoc ε, ε, τεχνικής ομάδας εργασίας για την εκπόνηση της συνθήκης ένταξης. Όλα αυτά είναι πολύ καλά νέα διότι δουλέψαμε σκληρά. Και προς το παρόν ο ισολογισμός αν θέλετε των διαπραγματεύσεων έχει ως εξή. Άνοιξαν 28 κεφάλαια και μέχρι στιγμής έχουν προσωρινά κλείσει 12, δηλαδή το 1 τρίτο του συνόλου των κεφαλαίων. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά από τα εκκρεμή κεφάλαια τα κεφάλαια 13 ε, αλία, 27 περιβάλλον, 31 εξωτερική πολιτική ασφάλεια και άμυνα μπορούν να ανοίξουν το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να ανοίξουμε και τα κεφάλαια αυτά και ελπίζουμε ότι και αυτά θα κλείσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι στόχος μας επίσης να επενδύσουμε ή μάλλον να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να κλείσουμε όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Η ε, Κροατία έχει ε, ολοκληρώσει το έργο της για τα πρόσθετα τέσσερα κεφάλαια και πολύ σύντομα θα κλείσει και τα επόμενα πέντε. Ε, καθόλου αυτό το διάστημα. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν απολύτως απαραίτητες για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι αναμένονται ακόμα πολλά. Ωστόσο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην νομοθετική ευθυγράμμιση με το κοινοτικό και κτημένο σε όλα τα κεφάλαια που άνοιξαν. Πρέπει να σας πω ότι το Κρατικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πάνω από 300 νόμους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη προσοχή έχει ε, δοθεί στην νομοθετική ευθυγράμμιση αν θέλετε, την εκπαίδευση και κατάρτιση εμπειρογνωμόνων, ως και προβλέπονται η διάθεση των ε, απαραίτητων κονδυλίων για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και λέω με απόλυτη πεποίθηση ότι η Κροατία επέδειξε την ικανότητα και την ετοιμότητά της σε όλα αυτά τα ευαίσθητα θέματα μεταρρυθμίσεων. Ε, Τούτο περιλαμβάνει και δύο τομεί πολύ σημαντικού, ναυπηγική και δικαστικό σώμα. Ω προ την ναυπηγική, κεφάλαιο 8. Η Κροατία συνεργάζεται στενά με τι υπηρεσίε τη Κομισιόν για να καθοριστούν οι συνθήκε για τον δεύτερο γύρο ε, ε, διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση έξι ε, ναυπηγείων. Σχετικά με το κεφάλαιο 23, δικαστικό σώμα και θεμελιώδη δικαιώματα αυξημένες προσπάθειες καταβάλλονται ώστε να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα αλλά και η αμεροληψία του δικαστικού σώματος. Τα τελευταία ε, λίγα χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ε, μείωση του αριθμού των ανεπίλητων ή ακρεμούντων δικαστικών υποθέσεων, τα οποία μειώθηκαν σε ε, ένα ποσοστό 8% ετησίως. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του 2005 ο αριθμός των εκκρεμούντων υποθέσεων ήταν 1,5 εκατομμύριο. Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι γύρω στους 860.000. Αυτή τη στιγμή... Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε την προσοχή μας στις τελευταίες 100.000 υποθέσεις που εκκρεμούν για παραπάνω από τρία χρόνια. Όσον αφορά την αξιολόγηση και τον διορισμό των δικαστών και των εισαγγελέων, λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλιστούν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Έτσι λοιπόν, για να βελτιώσουμε τη διαδικασία επιλογής, αυτή τη στιγμή ε, βρισκόμαστε στην τελική φάση της ίδρυσης μιας κρατικής σχολής. Εξορθολογισμός του δικτύου των δικαστηρίων βρίσκεται και αυτό σε καλό δρόμο με την εισαγωγή νέων μεθόδων και την εισαγωγή, εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα δικαστήρια. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι λαμβάνονται και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ε, εξουδετερώσουμε, να καταργήσουμε όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ώστε να αποκαταστήσουμε ένα δικαστικό σύστημα στα πρότυπα της Ευρώπης. Έχουμε προχωρήσει επίσης για την ενδυνάμωση της καταπολέμησης της ε, διαφθοράς. Υπάρχουν ε, ε, καλύτεροι συνονισμοί των ορμοδίων σωμάτων, καλύτερο νομικό πλαίσιο και αυτό οδήγησε σε περισσότερες επιτυχείς δράσεις. Ταυτόχρονα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της κατανόησης του κοινού για το πόσο βλαβερό και απαράδεκτο είναι το θέμα της διαφθοράς. Μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του διεθνούς ε, εγκλήματος προσθήθεμε να συνεχίσουμε με έντονη διεθνή συνεργασία και περιφερειακή, ε, αστυνομική και ε, δικαστική συνεργασία που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Η Κροατία αυτή τη στιγμή καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να ενδυναμώσει επίσης τις ε, διοικητικές της ικανότητες. Να Υπουργείο Διοίκησης έχει καθοριστεί και αυτό οδηγεί στον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης ε, γνώμη, με συμπληρωματική όρμη αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των γενικών διοικητικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. Θέματα στα οποία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να ε, πληρώσουμε τα κριτήρια benchmark της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να προετοιμάσουμε την Κροατία για τη μελλοντική της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μπορέσουμε να ωφεληθούμε κατά το μέγιστο από την ένταξή μας αυτή. Επίσης αναγνωρίζονται τα, οι προσπάθειές μας για την προστασία των μειονοτήτων και προσθέμεθα να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τομεί της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, στην αστυνομία και στο δικαστικό τομέα και τα ε, πολιτιστικά δικαιώματα και δικαιώματα στη της μειονότητας ιδίως των Ρώμα. Όσον αφορά το θέμα της επιστροφής των προσφύγων, αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσει 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα για να εξασφαλίσουμε την υποδομή, οικισμούς και να προωθήσουμε κοινωνικούς και οικονομικούς όρους για την καλή και αηφόρο επιστροφή. Η εφαρμογή του προγράμματος ε, της ε, ε, θεραπείας των κατοίκων είναι επίσης κάτι που προχωρούμε και θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε διμερή συνεργασία με τη Σερβία και τη Βοσνία Ρεσκοβίνη για να έχουμε ανταλλαγή των σημαντικών θεμάτων. Όσον αφορά το άνοιγμα του κεφαλαίου 23, εδώ σχετίζεται η συνεργασία μας στην ε, εξωτερική πολιτική. Εξακολουθούμε να είμαστε προσατημένοι στην πλήρη συνεργασία, στην νομένης και της πρόσβασης σε έγγραφα. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος ε, Ισαγγελέας Πράμας ε, επισκέφθηκε στο Ζάγκρεπ και μετά εγκατεδίθηκε μια ειδική μονάδα δράσης για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες προτάσεις του Ισαγγελέα. Η μονάδα αυτή έχει ήδη προετοιμάσει και υποβάλει στην εισαγγελία δύο έγγραφα εργασίας που αποτελούν τη βάση για μελλοντικές έρευνες. Ε, προ... Ετοιμάζεται περιττέρω πρόεδρος για τα τέλη της εβδομάδας. Εκτός από ε, υπάρχει μια ομάδα εμπρογραμμών που θα εξετάσει το θέμα αυτό για να μπορέσει η Task Force, αυτή η ομάδα κρούσης, να ολοκληρώσει την ερεύνα ικανοποιητικά όσον αφορά στις δράσεις που έχουν ανοιχθεί και την θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα benchmark του, του κεφαλαίου 23, η Κροατία ελπίζει ότι δεν θα υπάρχουν άλλα εμπόδια για το άνοιγμα αυτού του τόσο σημαντικού κεφαλαίου. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε πολύ καλά τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε κάθε τι που μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ε, την πλήρωση των ε, ε, προϋποθέσεων για την ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας αυτό κατά νου, θα συνεχίσουμε οι διαπραγματεύσεις με εμπιστοσύνη και ελπίζουμε ότι η κοινή μας εργασία θα είναι επιτυχής για να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέση του, μέσα του 2010. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ευρωπαϊκές ε, προσδοκίες των χωρών της ε, νοτιοανατολικής Ευρώπης βασιζόμενοι στην μεμονωμένη προσέγγιση και εκπληρώση των προβλεπωμένων κριτηρίων. Σε μια χώρα που έχει προχωρήσει περισσότερο στις διαπραγματεύσεις ένταξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κροατία υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία Ολοκλήρωση με την ε, Αλβανία, Βοσνία, Ορζεγοβίνη, Μοντενέγρο, Μακεδονία και Σερβία. Θα συνεχίσουμε να, να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με τους ε, γειτονές μας μέχρι να φτάσουν και εκείνοι στο στόχο της έλεγξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που ε, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από την ευρωπαϊκή προοπτική για την περιοχή αυτή. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Βοσνία γιατί αν ενδυναμωθεί η σταθερότητα της χώρας αυτής θα σταθεροποιηθεί ολόκληρη η περιοχή. Υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερα λειτουργόν κράτος με ξαφή ευρωπαϊκή προοπτική. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδικής Προεδρίας και τον ΗΠΑ που έχουν σαν στόχο πολιτική συνένεση μεταξύ όλων των ηγετών της Ευρώπης και εκείνων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Εξακολουθούμε να εξασφαλίζουμε ότι η Κροατία με αυξημένη συνεργασία σε όλους τους τομείς θα προωθήσει ιδίω τους τομείς ε, για την ενέργεια και την διαχείριση των υδατίνων πόρων. Η Κροατία μπορεί να είναι ένα παράδειγμα στις χώρες περιοχής στον, ε, στην οδό τους προς την Ευρώπη και θα ήθελα να πω ότι χαιρόμαστε μπορούμε να συμμεριζόμαστε τις ε, απόψεις και την εμπειρία μας με τους φίλους μας στις περιοχής. Κυρίες και κύριοι, η διαδικασία διάβρεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε και δίνει συνέχεια ε, εμπιστοσύνη, γνώσεις και πολλά κίνητρα για τη μεταρρύθμιση και συνεργασία προωθώντα έτσι σταθερότητα και νευμάρια στον Ήπειρό μας. Η Κροατία έχει προχωρήσει πολύ στη διαδικασία ένταξης τα τελευταία τέσσερα χρόνια και βρισκόμαστε κοντά στη τελική ευθεία. αυτά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις ενώπιόν μας και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την εργασία μας. Αυτή η ειδική προσέγγιση σε κύριους τομείς όπως η μεταρρύθμιση του κοστικού τομέα, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου κλίματος, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η δημιουργία διοικητικού μηχανισμού ικανού θα μας βοηθήσουν να ενταχθούν. Πολλά από τα κεφάλαια που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή είναι ακόμη πιο απαιτητικά υπό το φως της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που είναι όσοι μόνο σε εμά, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρο ότι θα είμαστε επιτυχεί σε αυτό το ιστορικό μα έργο και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μοιραστεί μαζί μα τι προσδοκίε και τον ενθουσιασμό μα. Οι διαπραγματεύσει τη Κροατία έχουν στρατηγική σημασία και σημαντική επίπτωση σταθερότητα για όλο το τομέα τη νότιο-ανατολική Ευρώπη, τη οποία το ευρωπαϊκό μέλλον στηρίζει απόλυτη η Κροατία. Η δική μα επιτυχία είναι η δική του επιτυχία. Και ένα τελευταίο σημαντικό σημείο. Η Κροατία χαιρετίζει θερμότατα την τελική υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας από τον Τσέχο Πρόεδρο και ε, το γεγονός ότι αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο θα τεθεί ε, σε ισχύ πολύ γρήγορα. Με την συνθήκη τη ανήγεινα ανοίγει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωση και έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι θα αναλυφθούν από όλους του οι ευθύνε και ε, ο ρόλος που πρέπει να παίξουμε στα πλαίσια της συνθήκης. Έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι η ορμή που έχει αποκτήσει η Κροατία πρόσφατα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του δημονισμού Ανοίγματο εκκλησίματο κεφαλαίων του επόμενου μήνε. Το να διατηρήσουμε την ορμή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το τόσο κρίσιμο, ε, κρίσιμο στάδιο στην διαδικασία ένταξης. Οι επιτυχίε της ε, ε είναι προ όφελο και της Κροατία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό πιστεύουμε απόλυτα ότι το κοινό μας έργο θα περάσει χωρίς προβλήματα από την τελική φάση και επαναλαμβάνω, ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια μέχρι τα μέσα του 2010. Τελειώνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά τη όργανα για όλε τι προσπάθειε και την ενίσχυση που μα προσέφεραν. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τόσο αξιόλογη υποστήριξή και το σκληρό έργο στην βοήθειά τους για μας κατά δια, ε, οδό αυτού του δύσκολου δρόμου. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τη δική σας υποστήριξη θα συνεχίσει η Κροατία στο δρόμο της και θα μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, να περάσουμε από κάθε εμπόδιο και να φτάσουμε εκεί που ανήκουμε δηλαδή στην κοινή μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σβόμποτα, ο οποίος ε, πήγε σε μια διήμερη επίσκεψη στην Κρατία και Σλοβενία. Κύριε Σλόμποτα, έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι αύριο θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μου, άρα λοιπόν δεν θα αφαιρέσω το χρόνο από άλλου συναδέλφου. Τρία σχόλια. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκομπονιάκ ε, για τις προσπάθειες που καταβάλει και για την ε, προσπάθεια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στη Σλοβενία είχα Είχα συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό κλπ. Ποτέ τα προηγούμενα χρόνια το κλίμα δεν ήταν τόσο καλό μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας όσο είναι τώρα. Οι άνθρωποι είχαν επικοινωνία, αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν ήταν καλό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τεράστιο ανοιχτό ε, παράθυρο ευκαιρίας ε, ώστε να προχωρήσει η συμμετοχή της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα θέμα ανοιχτό, τη διαδικασία επικύρωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε και με τις δύο αντιπολιτεύσεις ώστε να συμφωνήσουν ε, στην επικύρωση. Στην Κροατία είχα μία μακρά συζήτηση με τον πρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών, τον Ζόραν Μιλάνοβιτς και δούλεψα ώστε να δημιουργήσω τις απαραίτητες συνθήκες και για αυτόν και για αυτούς ώστε να συμφωνήσουν. Συνάδελφοι από το ΕΛΚ, ο κύριος Μπροκ και επίσης και άλλοι Γερμανοί θα πρέπει και αυτοί να καταβάλουν προσπάθεια ώστε να υποστηριχθεί η επικύρωση. Όπως είπα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Και τέλος, τρίτο σημείο και τελευταίο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής μας είπε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά ανοιχτά ζητήματα, αλλά είναι ζητήματα που μπορούν να επιληθούν πολύ γρήγορα. Και ιδιαίτερο ένα ζήτημα που είναι η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Έχω την εντύπωση ότι η Κροατία ενδιαφέρεται να αναβρεθούν όλα τα ντοκουμέντα, όλα τα έγγραφα. Ε, η ομάδα δράσης είναι κάτι πολύ καλό. Η ομάδα δράσης, το Task Force, θα πρέπει να υποστηριχθεί και από κάποιους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ενδεχομένως, ώστε να πιστεί και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες είναι, δεν έχουν πιστεί ακόμα ότι η Κροατία καταβάλει κάθε προσπάθεια. Θα το πω και στην έκθεσή μου αύριο. Η πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Κροατία αλλά και για τις άλλες χώρες και στην έκθεσή σας κύριε Πρόεδρε θα μπορούσατε να αναφέρετε όλες τις για, όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες ότι η συνεργασία με το Διεθνές δικαστήριο, Ποινικό Δικαστήριο είναι υψίστης σημασίας. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. Ο κύριος Πόσελτ και ο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τρεις υπογραφές άνοιξαν τον ε, δρόμο για την Κροασία, μία χθες στην Πράγα, δύο σήμερα στη Σουσχόλμη και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό και όπως ο συνάδελφος Σβόμποντα έτσι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Γι' αυτό θέλω να συμφωνήσω με την έγκλησή του προς τα πολιτικά κόμματα και στις δύο χώρες, και στη Σλοβενία και στη Κροατία, να εκμεταλλευτούν αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Και θα ήθελα να πω ότι αν δεν εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτό θα είναι εις βάρος όχι μόνο της Κροατίας αλλά και της Λοβενίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα. Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας πω όμως και κάτι άλλο. Ανησυχώ ιδιαίτερα μήπως στην τελευταία στιγμή υπάρξουν τεχνητά προβλήματα. Ε, ε, ευχαριστώ τον κύριο Βονάκ που αναφέρθηκε στα φυσικά εμπόδια που είναι αρκετά δύσκολα και που τα αντιμετωπίζει με μεγάλη ορμή. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως μήπως ε, κάποιες δυνάμεις ε, που κρυβόντουσαν πίσω από τα εμπόδια που τώρα έχουν ε, υπερβαθεί χρησιμοποιούν κάποια άλλα σημεία και θα να πω ότι το θέμα αυτό σύκτη, εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας, αλλά πώς προωθείται το σημείο αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Το λέω ξεκάθαρα. Είπαμε, κάθε χώρα θα πρέπει να ε, κριθεί βάσει των ικανοτήτων του. Και αν υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη ή ε, κάποιες πολιτικές δυνάμεις που θεωρούν ότι ε, θα πρέπει να συσχετιστεί με κάτι άλλο η ένταξη ε, της Κροατίας ένας ε, Γερμανός ανώτατος υπάλληλος ε, είπε πολύ άσχημα πράγματα σχετικά. Είπε βέβαια ότι είναι προσωπική του γνώμη, αλλά ας μην μας την παρουσίασε προσωπική του άποψη, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο διαπραγματευτή του κ. να μου πει κατά πόσο θεωρεί ότι είναι λογικό, αναμενόμενο να ανοίξουν όλα τα κεφάλαια μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτος για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους. Να συμβάλλουμε εμείς σαν κοινοβούλιο, αλλά στην τελευταία αυτή ευθεία να προσπαθήσουμε να επαγρυπνούμε να μην υπάρχουν τεχνητά εμπόδια. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει ο κύριος Στάλερ για δύο λεπτά. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε την πρόοδο της Κροατίας ε, στην οδό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό είναι καλό και για την Κροατία και για τους γείτονες της Κροατίας και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χάρηκα που ο εισηγητής κύριος Σφόποντα πήγε τη Δευτέρα στη Λιμπλιάνα γιατί έτσι μπόρεσε να δει πειραματικά ποια είναι η τελευταία πρόοδος της κυβερνήσης. Αυτό θα το βοηθήσει και για την εκθεσή του. Εγώ συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτή την ορμή που υπάρχει για να πετύχουμε την επικύρωση της συμφωνίας. Δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Στη Κροατία η Καθολική Εκκλησία εντάχθηκε κατά της συμφωνίας που είναι ασυνήθιστος η σημερινή πολιτική. Ε, διάφοροι επίσης διανοούμενοι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν μία ε, αναφορά κατά της ε, συμφωνίας. Στη Σλοβενία η κατάσταση είναι επίσης σαφής. Θα χρειαστούμε μία πλειοψηφία δύο τρίτων και θα πρέπει νομίζω να βοηθήσουμε να εξαλειφθεί το πρόβλημα αυτό μετά από 20 χρόνια. Στη Σλοβενία εμείς θέλουμε καλές συνθήκες γυτνίασης. η Κροατία να έχει ε, κατά νου και τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα των γειτόνων της. Έχω μια ερώτηση εδώ σχετικά. Προβλέπει κάτι αυτή τη στιγμή η Κροατία για να επιληθεί το πρόβλημα των συνόρων με την Βοσνία Ζεγοβίνη δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ενταχθούν οι χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα ήταν το πρόβλημα τεράστιο. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κάτσιν, δύο λεπτά. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Δρόβνακ, θα ήθελα να σας συγχαρώ και εσάς και την ε, κυβέρνησή σας και την επικεφαλή της που ε, διχθήκατε τόσο τολμηροί γιατί μόνο οι τολμηροί μπορούν να δημιουργήσουν ένα μέλλον καλύτερο από το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά κύριε Τρόγνετ έχω και κάποιες ανησυχίες. Οι δύο χώρες αποφάσισαν μονομερείς δράσεις μετά από την 25η εκ του 1909 ε, δεν θα πρέπει να προδικάζουν οτιδήποτε για τα σύνορα. Τώρα η δική σας πλευρά έκανε μια δήλωση μονομερή που θα ακολουθήσει μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ λογικό γιατί οι μονομερείς ε, δεν οδηγούν στο μέλλον. Και κύριε Ντρόγνα ελέγχθη ήδη ότι η δήλωση της διάσκεψης των επισκόπων είναι δυσνόητη. Πρόκειται για μια επίσημη ε, γνωμοδότηση. Δεν είναι κάτι που δηλώνει ένας επίσκοπος, αλλά όλη η Καθολική Εκκλησία στην Κροατία που λέει υπέρ της συνέχισης του βλοκαρίσματος και όχι για την υπογραφή της συμφωνίας. Έτσι λέει αυτή η συμφωνία. Τι έχετε να πείτε από αυτού Τελειώνοντας, έχω να σας πω ότι χαίρομαι που λέμε ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσει. Απ' την άλλη μεριά αναφέρονται κάποιες προθεσμίες που πάντα με ανησυχούν. Καλύτερο είναι να μην ορίζουμε προθεσμίες, αλλά να φροντίσουμε να υπάρχει μια συνοχή. Θα πρέπει η Κροατία να διαπραγματεύεται συνεχώς και να ε, προχωρεί συνεχώς. Αυτό είναι που θέλουμε και μου μας ε, ενώνει. Και τέλος, στρεφόμενος προς τον συνάδελφο Σβόμποντα, έχω να πω ότι ο, ο κόσμος δεν είναι μαύρο-άσπρος, ούτε η πολιτική είναι κόκκινη και μαύρη, υπάρχει και κίτρινο και πράσινο. Όλος ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να φροντίσει ούτως ως η Κροατία να επικυρώσει τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Το λόγο είναι συνάδελφος Βάγκνερ. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Καταρχήν έχω να πω ότι και εμείς χαιρόμαστε σαν πολιτική ομάδα για την καλή πρόεδρο που επετέλεσε η Κροατία το παρασπένο έτος. Αλλά όσον αφορά το δικαστικό τομέα είναι πολύ επικριτική η έκθεση της Κομισιόν οργανωμένο έγκλημα, επιστροφή των προσφύγων κλπ. Σημεριζόμαστε τις ε, ανησυχίε αυτές και τι κριτικέ. και θέλω να μου πείτε πώ θέλετε να αποθετήσετε του ε, τομείς Επίσης, ε, τον Μάρτιο του 2009 η οργάνωση Φέλη ε, της Γης ε, Friends of the Earth Κρέτσια έκανε μια διαδήλωση γιατί η σχετική νομοθεσία δεν προωθείται επαρκώς η νομοθεσία για το περιβάλλον. Τώρα η κυβέρνηση είπε ότι θα επιβάλλει στην μη κυβερνητική οργάνωση αυτή ε, κυρώσεις γιατί υποτίθεται ότι μόλυναν την πόλη όταν έκανα μια διαδήλωση και θα φτάσουν μέχρι τις 100.000 ε, ευρώ. Εσείς μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι στην ε, δικαστική αυτή υπόθεση κατά των φίλων της γης, των Friends of the Earth, θα κτηρηθεί κάποιο μέτρο. Σας ευχαριστώ για την ε, απάντησή σας. Τώρα τα είπα γερμανικά και ο κύριος Πρόπ έχει φύγει. Ευχαριστώ. Το λόγος της συνάδελφου Ιμπρίζα Ζιτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ. Χαίρομαι που έχουμε ένα καλό διάλογο. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση να σας υποβάλω. Αναμένετε αυτό το άρθρο, το κεφάλαιο συγγνώμη 31 να μπλοκαριστεί που αφορά τις εξωτερικές σχέσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, η οποία είναι σημαντική ε, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή. Και η περίπτωσή σας νομίζω ότι δείχνει τη σημασία των προβλημάτων και την επίλυσή τους για την ένταξη, γιατί ακόμα και αν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε στα κείμενα ότι τα προβλήματα που αφορούν σχέσεις καλής γειτονίας δεν πρέπει να εμποδίζουν, στην πράξη όλοι ξέρουμε ότι εμποδίζουν. Άρα η περίπτωση Κροατίας είναι πάρα πάρα πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο η παρέμβαση του Επιτρόπου Ρεν βοήθησε στην επίτευξη της, Συμφωνίας και κατά ποιο τρόπο ε, θέλοντας με αυτό να ρωτήσω αν πραγματικά η παρέμβαση της Επιτροπής σε υπάρχοντα θέματα στα Βαλκάνια μπορεί πραγματικά να δώσει διεξόδους. Ευχαριστώ. Με την παρέμβαση της κυρίας Πακ για δύο λεπτά θα κλείσουμε την χειροτονέλη Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Χόριαξ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας που κατέληξε πού βρίσκονται τα προβλήματα και τι έχετε καταφέρει μέχρι στιγμή. Συγχαρητήρια. Θα περιοριστώ σε δύο σημεία μόνο. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα Σλοβενίας-Κροατίας προφανώς μπορεί τώρα να επιληθεί. Εάν σε κάθε χώρα ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί. Ο κύριος Φόμποντα είπε ότι θα άσκηση επίση στην ε, αντιπολίτευση στην Κροατία, ε, γιατί μέχρι στιγμή δεν ε, τοποθετήθηκε. Μάλιστα, ο υποψήφιο για την Προεδρία καταψήφισε. Δεν ξέρω κατά πόσον εγώ μπορώ να έχω την ίδια επίδραση στους Σλοβαίνους συναδέλφους μου στη Σλοβενία. Θα προσπαθήσω όμως να πείσω και άλλους για να το καταφέρουμε αυτό. Ε, θα πρέπει τώρα να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και Θα ήθελα να πω και προς τον κύριο Καλά και εγώ θα ήθελα να μου πει ο ήμουν στο Μαυροβούνιο, τι γίνεται με τα προβλήματα των συνόρων της Κροατίας και του Μαυροβουνίου, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, λύνονται, δεν υπάρχουν και επίσης το ίδιο για το πρόβλημα για τη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Αλλά ξέρω κύριε λέω ότι ακόμα και αν δεν επιληθούν, δεν θα κάνει η Κροατία το ίδιο που έκανε αυτή τη στιγμή που είδε με την Σλοβενία. Δεν θα κάνει στους άλλους αυτό που τους έκανε εκείνη. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα νομίζω. Εδώ που θέλω να ταχθώ είναι στο γεγονό ότι η καθολική διάσκεψη των επισκόπων ανακα... αναμίχθηκε σε αυτό το θέμα. Εγώ είμαι καθολική. Προσπαθώ πάντα να στηρίξω την Εκκλησία, αλλά μου φαίνεται πραγματικά ανήθικο να αναμειγνύονται σε κάτι τέτοιο. Ποιον καλύπτουν. Δεν είμαι σίγουρη ότι οι επίσκοποι ξέρουν ακριβώς τι λέει αυτό το κείμενο. κάποιος που έχει προσβληθεί νομίζω ε, θεωρεί ότι δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη στη συζήτηση αυτός έχει αναδαβλήσει αυτή την κατάσταση ο νοήτο εγώ θα ήθελα ρητά να πω ότι πραγματικά η Καθολική Εκκλησία δεν πρέπει εδώ να αναμειχθεί όπως και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιτρέπεται να αναμειχθεί στην πολιτική στο στη Σερβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πακ. Ο αρχηγός της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει το λόγο για τις πρώτες απαντήσεις. Υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων. Ας αρχίσω με αυτό σχετικά με τις σχέσεις Κροατίας-Σλοβενίας. Θα είμαι πολύ σύντομος. σημερινή μέρα είναι μια πολύ καλή ημέρα για τις σχέσεις Κροατίας-Σλοβενίας. Και ε, θα κατανοήσετε για ποιο λόγο δεν θα κάνω κανένα άλλο σχόλιο επ' αυτού από το βήμα αυτό. Διότι σήμερα οι δύο πρωθυπουργοί μας ομίλησαν στην Στοκχόλμη και μίλησαν σοφά τα λόγια τους έχουν πολύ σημαντικά μηνύματα και νομίζω ότι σήμερα δεν πρέπει να προσθεθεί τίποτε άλλο ε, ασφαλώς δε, πολύ περισσότερο δε από έναν δημόσιο υπάλληλο όπως είμαι εγώ. Άλλο ερώτημα. Μπορούμε να, να ανοίξουμε όλα τα κεφάλαια μέχρι το τέλος του έτους. Υπάρχουν ακόμα πέντε κεφάλαια που πρέπει να ανοίξουν. Τα 13, 27 και 31 για τα τρία αυτά σας μίλησα ήδη. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Η διαπραγματευτική μας θέση έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και καιρό. Είναι τεχνικά έτοιμα τα κεφάλαια αυτά για συζήτηση στην ομάδα και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει και η Σλοβενία μπορούν αυτά τα κεφάλαια να ανοίξουν τις προσεχείς ημέρες ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ακόμα μια διακυβερνητική υποσχεδική προεδρίας. Το κεφάλαιο 8. Πολιτική ανταγωνισμού. Εκεί υπάρχουν διάφοροι στοχοδείκτες, τους ε, έχουμε καλύψει όλους, αλλά υπάρχει ένα σχετικά με τα ναυπηγεία, όπου θα πρέπει εμείς πρώτα να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ιδιωτικοποίησεων. Ήδη κάναμε τον πρώτο γύρο. Είμαστε σε στενή επαφή με την Κομισιόν, που βοήθησε πολύ με τις διαβουλεύσεις που είχαμε μαζί της. Η διαπραγματευτική μας θέση είναι έτοιμη να υποβληθεί. Είμαι βέβαιος ότι και αυτό το κεφάλαιο μπορεί να ανοίξει το Δεκέμβριο. Το κεφάλαιο 23. Εξα, εξαρτάται από το τι θα πει ο ε, Γενικός Εισαγγελέας ο Μπράμιτς. Ελπίζουμε ότι η γνωμοδότηση θα είναι θετική. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να, να ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο. Διότι τρία επίσημα τρει επίσημοι στόχοδείκτε, το ένα για το δικαστικό στόμα, το άλλο για την καταπολέμηση τη διαφθορά και το τρίτο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τα τρει αυτοί στοχοδείκτε έχουν καλυφθεί από την Κροατία και έχουμε ένα πολύ θετικό σχόλιο από την Κομισιόν. Αλλά όπως προβλέπουν οι κανονισμοί θα πρέπει να επαληθευτεί αυτή η επίσημη άποψη της Κομισιόν να ε, επαληθευτεί από τις χώρες μέλη. Θέμα συνόρων. με τη Βοσνία, Ζεγοβίνη, τη Σελβία και το Μαυροβούνιο. Ας αρχίσω με το Μαυροβούνιο. Ναι, αφορά τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη τελική συμφωνία. Ε, για να φέρουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο. Και νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης των ζητημάτων υπό διεθνή διατησία. Σερβία, Βοσνία, Ερζεγοβία. Υπάρχει θετική προσέγγιση για να εντατικοποιηθεί ο διάλογος. Προσεγγίσαμε τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και διμερός σχετικά με τα σημεία διέλευσης ε, εξαιτία του κεφαλαίου 24. Και επειδή αυτά θα καταστούν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ γρήγορα. Πρέπει λοιπόν να διαπραγματευτούμε κάποια θέματα σχετικά με την ταξινόμηση των συνόρων κλπ. Είμαστε ανοιχτοί για να ενισχύσουμε τον διάλογο αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι ο διάλογος αυτός θα αποδώσει καρπούς. Και τα θέματα θα επιληθούν. Και δεν βλέπω να υπάρχει κανένα εμπόδιο που να μην μπορούμε να διαπραγματευτούμε. When it comes to Έρχομαι τώρα στην οργάνωση Friends of the Earth. Εγώ ως επικεφαλής διαπραγματευτής θα μπορώ να σας εγγυηθώ ότι κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε οι Friends of the Earth, οι φίλοι της γης, να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο πρέσβης ε, Μπρίσοβιτς μου, δίνει, μου έδωσε ένα σημείωμα που λέει ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται αλλά το ερώτημά σας κατεγράφει και θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή όταν επιστρέψω στο Ζάγκρεπ. Προσωπικά θα ασχοληθώ Μείνετε ήσυχο η ανησυχία σα θα ληφθεί υπόψη. Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε στο κεφάλαιο 31. Κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δεν έχει ανοίξει ούτε έχει κλείσει. Κροατία είναι της άποψης ότι εφόσον το ζήτημα με τους Σλοβαίνους φίλους βρίσκεται σε καλό δρόμο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προχωρήσει γρήγορα και αυτό το κεφάλαιο. Πιστεύουμε ότι η Κροατία έχει πολύ καλές επιδόσεις από την αρχή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, διότι αμέσως γίναμε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό μιλάει από μόνο του για την ετοιμότητά μας στον τομέα της κοινή άμυνας και ασφάλειας. Η Κροατία αυτή τη στιγμή είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, φέρνει και υποστηρίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο. Η Κροατία σταθερά συμμορφώνεται σε όλα τα διεθνή φόρα με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια. Η Κροάτης διπλωμάτης είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας και λοιπά. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν την ετοιμότητα και την δέσμευση της Κροατίας ε, να δεχθεί όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την κοινή εξωτερική ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Εφόσον λοιπόν λυθεί το ζήτημα με τη Σλοβενία, πιστεύω και είμαστε στο δρόμο για να ανεβρεθεί αυτή η λύση, τότε είμαι βέβαιος ότι να προχωρήσω πολύ γρήγορα και το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει κανένα ερώτημα που δεν απάντησα. Α, ναι. Ε, Επίτροπος Ρεν. Πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Επιτρόπου. Ασφαλώς ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος υπό δυσχερείς συνθήκες επένδυσε πολύ προσωπική προσπάθεια. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι ο δικός του ρόλος είναι σημαντικός στο να επιμείνει σε αυτό το πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ε, χάρη στο σύστημα των benchmarks, των στόχοδικτών, προχώρησε αυτό το πολύ ακαθόδες ζήτημα. Χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση υποψήφια για ένταξη χώρα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει και γι' αυτό πρέπει να πω ότι η Κομισιόν βοήθησε πολύ, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των εγγράφων. Και είναι δύσκολο όχι μόνο για μας που είμαστε υποψήφια χώρα, αλλά και για την ίδια την Κομισιόν και για τις άλλες χώρες μέλη. Πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να σας πω τον τεράστιο όγκο των εγγράφων. Χιλιάδες έγγραφα. Ναι, όλη η ΡΕΝ διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δεν το έπρατε, δεν θα είχαμε προχωρήσει όσο έχουμε προχωρήσει σήμερα. Και νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κουκαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω ερωτήσεις. Έχω τρεις σύντομες θετικές γενικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντρόγκαν, για την πληροφορίες σας. Χάρηκα που η δική σας αξιολόγηση για την Κροματεία συμπίπτει με την αξιολόγηση της έκθεσης πρόοδου. Η έκθεση πρόοδου λέει πραγματικά ότι υπάρχει μια συνεχής πρόοδος. Το συνεχής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι όλοι αναμένουμε στο μέλλον να δούμε να συνεχίζεται αυτή η συνεχής πρόοδος. Όπως είπε ο κύριος Προσφόποντα, πολλά πρέπει να ε, γίνουν ακόμα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γιατί μέχρι στιγμής προχωράτε πολύ καλά. Και όλοι θα περιμένουν να συνεχίσετε έτσι και στο μέλλον. Και μην περιμένετε ότι θα σας κάνουμε καμιά έκπτωση ή καμιά χάρη. Τον εναντίον θα πρέπει να συνεχίσει τις σκληρές σας προσπάθειες για να φτάσετε εκεί που πρέπει. Δεύτερη παρατήρηση. Η θετική εξέλιξη της δικασίας ένταξης της Κροατίας έχει σημαντικές θετικές επικοδομητικές επιπτώσεις στις άλλες χώρες της περιοχής. Το είπατε, αλλά θέλω να το τονίσω. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σαν περισσότερη πολιτική ευθύνη για σας, γιατί όλοι θα σας παρακολουθούν και θα κρίνουν τις μελλοντικές δυνατότητες έναξης της περιοχής σύμφωνα με τις δικές σας ε, αποδόσεις. Και θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με ε, τη χώρα, για τη χώρα μου την Σλοβακία είναι ιδιαίτερα ευχαριστώ όπου η χώρα σας προχωράει τόσο καλά. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Κούχαν. Η κυρία Μπότσκουρτ. Α, αναπληρώτρια. Η κυρία Γιαννάκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να συγχαρώ τον εκπρόσωπο της Κροατίας για όσα μας περιέγραψε και για τις προσπάθειες. Εγώ ήθελα να κάνω δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά στο ζήτημα των προσφύγων. Αν δηλαδή, το έφυξε και η κυρία Πακ προηγουμένως, αν δηλαδή υπάρχει κάποια ελπίδα, γιατί όσο περνά ο χρόνος βέβαια οι άνθρωποι μονιμοποιούνται εκεί που έχουν καταφύγει, αν υπάρχει κάποια ελπίδα για την πραγματική ανταλλαγή προσφύγων μεταξύ Βοσνίας Αζεγοβίνης και Κροατίας. Και το δεύτερο ζήτημα, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ε, σχετικά με τη συμφωνία με τη Σλοβενία. Ε, θεωρεί ο εκπρόσωπος της Κροατίας ότι ε, οι διαμαρτυρίες που υπάρχουν εντός της Κροατίας για το θέμα αυτό μπορούν να δημιουργήσουν κάποιους, κάποιες τριβές και εθνικιστικές αιτιάσεις λόγω του καθορισμού των συνόρων που πιθανόν θεωρείται μέσα στην Κροατία ότι είναι εις βάρος της Κροατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου. Η κυρία Μπότσκουρτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είχα μία ερώτηση για να δώσω συνέχεια σε αυτό που ακούστηκε κατά τη συζήτηση, δηλαδή η ελπίδα ότι θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα κεφάλαια το συντομότερο δυνατό. Αναρωτιέμαι όμως, επειδή στο κείμενο της Κομισιόν αναφέρεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία, εάν ε, δεν θα ήταν καλό να μην κοιτάμε μόνο τις ημερομηνίες και τη λήξη προθεσμιών αλλά και τα αποτελέσματα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς πού βασίζεται όλη αυτή η πεποίθηση ότι τα 2010 θα έχουν τελειώσει τα πάντα σε happy end. Ο κύριος Βάγκελ για δύο λεπτά είναι ο σκιώδης εισηγητής της Άλτε. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Λέχθη ότι μπορούμε σήμερα να είμαστε πιο ενθουσιώδεις γιατί δύο τολμηροί πρωθυπουργοί υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα περαιτέρω βήματα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έργο μας. Η διαδικασία επικύρωσης και ενδεχόμενα εμπόδια στην οδό για την αποδοχή του θέματος και στη Σλοβενία και στην Κροαστία ε, είναι αρκετή πολύπλοκη. Θα χρειαστεί λοιπόν μια πολιτική ευαισθησία για να μην θριαβολογούμε πολύ έγκαιρα, πολύ νωρίς, γιατί λέμε ότι ο θρίαμβος του μεν είναι η αποτυχία του δε. Αυτό δεν είναι καλό αυτή η ιστορία με την Κροατία, μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας δηλαδή, για τα σύνορα, κατέδειξε ότι το θέμα των σύνορων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέματα σύνορων είναι θέματα πάντα που ξεπερνάνε τα διμερή συμφέροντα. Και χώρε που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα έγκαιρα ε, κατά δυνατόν πριν ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να πω ότι η έκθεση του συναδέλφου Σόμποντα, που θα εξετάσουμε αναλυτικά αύριο, ανοίγει πολλά ερωτήματα για την Κροατία. Η Κροατία τα γνωρίζει όμω αυτά και τη εύχομαι κάθε επιτυχία και κάθε τύχη στην περιττέρου τη οδό. Για δύο λεπτά ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να, να θέσω δύο ερωτήματα στον ε, κύριο Υπουργό από την Κροατία. Πριν το κάνω αυτό, θα ήθελα ε, να του πω ότι του εύχομαι η χώρα του να μην εισπράξει κάποτε, όπως η Ελλάδα, από επίσημους Ευρωπαϊκής Ένωσης την έκφραση «The game is over». Το λέω αυτό διότι, όπως θα ξέρει πολύ καλά ο κ. Υπουργό, μπαίνει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τους κανόνες του παιχνιδιού τους, κανονίζει το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλες πολυεθνικές και ελπίζω και εύχομαι ε, ο λαός της ε, Κροατίας να μην το μετανιώσει. Επίσης, ε, εύχομαι στο μέλλον και ο λαός της Κροατίας να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να αποφαίνεται με δημοψήφισμα για σημαντικές αποφάσεις και στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα μου πει ο κύριο Υπουργό είναι ζητήματα τη Κροατία. Να περάσω τώρα να γίνω κάπω πιο συγκεκριμένο. Πρώτον, ε, και στην έκθεση πρόοδου, αλλά και σήμερα έγινε λόγο για τα προβλήματα τη Κροατία με το Διεθνέ Δικαστήριο τη ε, Χάγη για την πρώην Οικοσλαβία. Αυτό σημαίνει ότι η Κροατία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει αυτό το δικαστήριο. Καλά θα κάνει να μην το αναγνωρίσει. Εγώ λέω ότι είναι παράνομο και καλά κάνει η Κροατία και δεν το αναγνωρίζει. Εγώ θέτω αυτό το ερώτημα όμως. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να θέσω και τελειώνω είναι το εξή. Αύριο θα δούμε μια έκθεση προόδου ε, και της χώρας του όσον αφορά την ε, ενταξιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ε, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξέρετε πάντα θα με ενδιέφερε και η γνώμη των χωρών για τις, εκθέσει εκθέσεις πρόοδου αυτές. Παραδείγματος χάρη γίνεται λόγος, προχώρησε στον τάδε τομέα, δεν προχώρησε στον άλλον τομέα κτλ. Είναι πάντα η άποψη του εισηγητού. Θα είχε ένα ενδιαφέρον όμως να ξέρουμε και ποια είναι και η γνώμη των χωρών που τους αφορούν οι συγκεκριμένες εκθέσεις. Δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχουν δυσκολίες. Και θα ήθελα, επειδή δεν πρόκειται να έχουμε με τους άλλου ε, με τις άλλες χώρες εκπροσώπους των χωρών τους. Θα ήθελα εντελώς επιγραμματικά, αν ο κύριος Υπουργό είχε την καλοσύνη, σε ορισμένα δύο-τρία σημεία βασικά, να μας πει ποιες είναι οι δυσκολίες της Κροατίας στο να εκπληρώσει ορισμένους από αυτούς τους στόχους που τίθεται ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. η συνάδελφος Παζό από τη Λίμπε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε ήδη από τους προλήσαντες πολλά ενδιαφέροντα και θα ήθελα να χαιρετήσω την πολιτική τόλμη των χωρών που υπέγραψαν σήμερα την Συμφωνία Διατησίας. Αυτό είναι η πρώτη σοβαρή συμφωνία μετά το 2001. Και ελπίζω ότι οι βουλευτέ και των δύο χωρών θα τολμήσουν να επικυρώσουν μέχρι το Δεκέμβριο έγκαιρα. Καταλαβαίνω τι ε, επιφυλάξεις σας ε, και καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να επισέλθετε στις λεπτομέρειες της ε, συμφωνίας αυτής για την διαδικασία διατησίας, μια που μόλις σήμερα υπεγράφει. Θα με ενδιαφέρε όμως η Κροατία ποιον θα ορίσει σαν διαιτητή σε αυτή την ομάδα. Και θα ήθελα να υποβάλω και μια ερώτηση που δεν υπευλήθη ακόμα σήμερα και σχετίζεται με την έκθεση πρόοδου για την Κροατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο άρθρο, για τις, στο κεφάλαιο συγγνώμη, για τη σχέση μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος για την Μπάνκα Λουμπλιάνσκα και με τις αποταμιεύσεις ε, Κροατών αποταμιευτών. Πολλά διαβάζουμε γι' αυτό, αλλά σας ρωτάω τι είναι η δική σας γνώμη. Ε, Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Λοιπόν, τελική απάντηση. Το πρώτο θέμα νομίζω έχει να κάνει με το ζήτημα των προσφύγων. Να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δική μας θέση σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι αναμφισβήτητο ότι για μας η επιστροφή και ενσωμάτωση των προσφύγων είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Ήδη ανέφερα ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σχετικά με τους προσφύγους πρόσφυγες και τους εσωτερικούς εκτοπιστέντες. Μέχρι στιγμής 221.000 εκτοπιστέντες επέστρεψαν και 126.000 πρόσφυγες επέστρεψαν και όπως είπα επενδύσαμε 5,3 δις ευρώ περίπου από την πρώτη ημέρα για ανασυγκρότηση ε, ανοικοδόμηση για να σας δείξω την κλίμακα της προσπάθειάς μας 146.000 σπίτια ανακατασκευάστηκαν Είμαστε της άποψης ότι εκπληρώσαμε τις υποχρεώσεις μας ε, με βάση την δήλωση του Σεράγεβο του 2005 και επιπροσθέτως για να διευκολύνουμε την επιστροφή ε, όλων η Κροατία εφαρμόζει ένα πρόγραμμα δράσης, ειδικό πρόγραμμα δράσης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η στενότητα, η οικονομική στενότητα καθιστά το ζήτημα κάπως πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά παρά τα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε με όλη μας την προσπάθεια, με όλη μας τη δύναμη την προσπάθεια. Ένα άλλο ζήτημα και ελπίζω να έχετε Ακόμα ένα λεπτό υπομονής. Πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την προσπάθεια που καταβάλει η χώρα. Οι φίλοι μας στη Σερβία αυτή τη στιγμή λένε ότι περίπου 70.000 πρόσφυγες από την Κροατία ζουν στη Σερβία. Κατά τη γνώμη μας, τα στοιχεία αυτά έχουν υπολογιστεί έτσι πολύ αυτόματα και θεωρούνται δεδομένα από κάποιους, χωρίς να τεκμηριώνονται. Η έκθεση πρόοδου του 2009 αναφέρει ότι περίπου 80.000 Σέρβοι είναι εγγεγραμμένοι ως πρόσφυγες. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της, είπα, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Ε, δεν υπερβαίνουν τις 25.000. Πολλοί άλλοι έχουν αποκτήσει τη σελβική υπηκότητα. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Τα σχόλιά μου δεν στρέφονται εναντίον του δικαιώματος του οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε θέλει να επιστρέψει. Οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί να επιστρέψει. Ωστόσο, χρειάζεται να υπάρξει μια σαφή θέση από σερβικής πλευράς διότι στα τελευταία ανάλυση έχουν περάσει και 18 χρόνια. Σας διαβεβαιώ ότι στο ζήτημα των προσφύγων θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ό,τι απαιτείται γιατί θεωρούμε ότι όχι μόνο είναι η υποχρέωσή μας στο πλαίσιο της ενταξιακής ε, διαδικασίας αλλά και υποχρέωσή μας ως ε, χώρας η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2010 θέλουμε να πετύχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, προσωρινά να κλείσουμε όλα τα κεφάλαια και δεύτερον, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε και τη συνθήκη ένταξης. Μετά θα αρχίσει βέβαια η διαδικασία επικύρωσης. Από πλευρά μας είναι εξαιρετικά δύσκολη δουλειά, αλλά έχουμε ε, την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών μελών. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο. Από το 1992 ασχολούμαι με την ε, διπλωματία της χώρας μου και ξέρω ότι δεν είναι ε, καθόλου εύκολο. Διεθνές ποινικό δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Η Κροατία συνεργάζεται στενά. Η Κροατία από την σύσταση του δικαστηρίου αυτού έλαβε 848 αιτήματα για αρρωγή προς τον ε, Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και εμείς απαντήσαμε 847 ε, και μισό. Και ε, σε ένα εξ αυτών απλώς ε, εκρεμεί η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα. Σας περιέγραψα ακριβώς και με λεπτομέρειες τι ακριβώς κάνουμε, δεν θα επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες. Κυρία μου, η ερώτησή σας αφορούσε στο ποιος θα είναι ο διαιτητής από πλευράς της Κροατίας. Εν πάση περιπτώσει όμως θα είναι ένας διετής εμπειρογνώμων. Αυτός ο ανανεωμένος διάλογος με την νέα δυναμική και τον αμοιβαίο σεβασμό δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ένα πρόβλημα πάρα πολύ σύνθετο, δημιουργεί λοιπόν το κατάλληλο περιβάλλον για την επίλυσή του. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Ε, ναι, μιλήσατε για τις δυσκολίες της διαδικασίας. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Απλώς θα ήθελα να αναφέρω κάποια κεφάλαια τα οποία για μας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Κάθε κεφάλαιο έχει τη δική του σημασία, αλλά για μας, εκτός από το κεφάλαιο 23, ε, στο οποίο αναφέρθηκα επί μακρόν, υπάρχει και το κεφάλαιο 22, περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά ταμεία. Εκεί πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική μας ικανότητα. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Εστιάζουμε την προσοχή μας εδώ ιδιαίτερος. Στόχος μας στη φάση αυτή δεν είναι μόνο να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις, αλλά επίσης ταυτόχρονα να δημιουργούμε τις απαραίτητες διοικητικές δομές που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους μετά την ένταξη. Την ενταξιακή μας διαδικασία δεν τη βλέπουμε ως αυτό σκοπό. Ε, ο βασικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ενισχύσουμε τις δυνατότητες και ικανότητες της Κροατίας σε όλους τους τομείς για να αποδείξουμε ότι πραγματικά είμαστε ένα άξιο μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Molto bene. Πολύ ωραία συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ. Πολύ εγκάρδια συνάντηση και ενδιαφέρουσα, στην οποία συμμετείχαν πολλοί άριθμοι συνάδελφοι. Ο μιλητής μας απάντησε με πολύ ακρίβεια, ελπίζω όλη αυτή η διαδικασία, εύχομαι δηλαδή να πάνε όλα καλά. Μια ένα σύντομο τεχνικό διάλειμμα και στις 6 θα συνεχίσουμε με τα επόμενα σημεία στην ημερήσια διάταξη. <laughs>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 Colleghi, visto che siete quasi... Συνάδελφοι, επειδή είμαστε ίδιοι, μπορούμε να μειώσουμε για τεχνικούς λόγους το διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το σημείο που αφορά στην πρόταση ψηφίσματος για τη στρατηγική διεύρυνθης για 2009 Δυτικά Βαλκάνια, Ισλανδία και Τουρκία. Να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που είμαι εισηγητής έστω και αν ο ρόλος μου δηλαδή είναι καθαρά τυπικός γιατί η πραγματική δουλειά και η ουσία αυτού του κειμένου οφείλεται κυρίως στους συναδέλφους που θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και οι οποίοι συνάδελφοι ε, είναι αυτοί που ε, είχαν το διάλογο με τις χώρες που θα γίνουν μέλη και εύχομαι, τους ευχαριστώ δηλαδή, και εύχομαι να μπορέσουν να εμψυχώσουν όλη αυτή τη συνάντηση και να τονίσουν ποια είναι και τα καυτά σημεία όλων αυτών των θεματικών. Τώρα, γιατί τόσο γρήγορα αρχίζουμε να ασχολούμεθα με αυτό το ψήφισμα. Μα γιατί θα πρέπει πριν εκφραστεί το Συμβούλιο να δώσουμε και εμείς τον προσανατολισμό μας για αυτά τα θέματα. Θέλουμε εμείς να τροφοδοτήσουμε την όλη συζήτηση που ξεκίνησε η Κομισιόν για τη στρατηγική της διεύρυνσης και να είμαστε παρόντες όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι το τέλος, δηλαδή τη στιγμή της λήψης της απόφασης. Ε, η διαδρομή της διεύρυνσης ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, κυρίως στα ανατολικά σύνορα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το ότι συνέβη τα τελευταία χρόνια, έστω και να έχουμε δυσκολίες, είχαμε και δυσκολίες στο να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε χώρες οι οποίες μόνο πρόσφατα γνώρισαν τη δημοκρατία. Ακόμη βέβαια δεν πετύ, το πετύχαμε, αλλά από το 2003 και μετά τα οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θεωρήθηκαν ότι έχουν ευρωπαϊκή χρειά. Ε, δύο μεταξύ αυτών, έναν τον ακούσαμε προηγουμένως, δηλαδή η Κροατία και η πρώην ε, Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ε, και η Ισλανδία η οποία αντιμετώπισε ε, την ε, τεράστιες επιπτώσεις της κρίσης θέλει να γίνει μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς και το είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε ότι κατάφεραν να τα βρούνε οι Κροάτες με τους Σλοβαίνους για το θέμα των συνόρων και αυτό έδωσε μια σημαντική όθηση στο να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εμείς λοιπόν ε, έχουμε εμπιστοσύνη, το ακούσαμε δηλαδή και από τον ε, αρχηγό της ε, αντιπροσωπείας διαπραγματεύσεων της Κροατίας ότι θα είναι σύντομα έτοιμη και οι επιτυχίες της ΦΥΡΟΜ είναι πολύ σημαντικές οι διαπραγματεύσεις ε, θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο και το θέμα του ονόματος επίσης θα πρέπει να λυθεί εγκαίρως. Έχουμε καλά στοιχεία τώρα στα χέρια μας για να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα, θα συμβεί. Τώρα για τη Βοσνία τα πράγματα δεν είναι και τόσο ικανοποιητικά. Ο διάλογος ε, για τις ε, θεσμικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστεί αλλά και σε αυτό έχουμε καλές ε, δυνατότητες ούτως ώστε οι πραγματεύσεις να προχωρήσουν θετικά. Η Τουρκία, η Τουρκία έχει ακόμη πολλές δυνατότητες για να προοδεύσει ας πούμε συμφωνία με την Αρμενία που έχει αρχίσει και τελειοποιείται και είχαμε και ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα αλλά ακόμα έχει πολλή δουλειά κυρίως ε, στα θέματα ελευθερίας της έκφρασης και ελευθερίας του θρησκεύματος. Αλλά υπήρξαν και μερικές πρόοδοι. Τώρα, για τις άλλες ε, χώρες, Μαυροβούνιο και Αλβανία, και αυτές βρίσκονται στο σωστό δρόμο, πρέπει να συνεχίσουν με τις μεταρρυθμίσεις. Και η πρόσφατη απόφαση που λάβαμε για τις ε, θεωρήσεις, για τις βίζες, ενθαρρύνει όλη αυτή τη διαδικασία. Για τη Σερβία το ενδιάμεσο πρωτόκολλο θα πρέπει να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατό. Εγώ περιορίστηκα απλώς εδώ να κάνω μία παρουσίαση με τίτλους, διότι όπως έλεγα και στην αρχή, όλη αυτή τη δουλειά την έκανε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων με τεράστια εμπειρία και γνώση στον τομέα αυτό και σε αυτούς λοιπόν θα αφήσω ε, την ε, πρωτοβουλία για να αναλύσουν τα διάφορα θέματα. Η κυρία Πάκα έχει πρώτη το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις περιπτώσεις. Νομίζω Όσον αφορά στο παράγραφο 12 Σερβίας, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Σερβία καλύτερα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα ως προς τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Τοπικές εκλογές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο στο Κωσυφοπέδιο και το Βελιγράδι ε, ε, έκανε έκκληση προς τους Σέρβους να συμμετάσχουν σε εκλογές αυτό. Θέλουμε να έχουν μια νέα προσέγγιση και ίσως θα έπρεπε και εμείς να βοηθήσουμε. Έχω μια τροπολογία για αυτή τη συγκεκριμένη παράγραφο την οποία θα υποβάλω αύριο. Δεύτερον, στο, στην παράγραφο 13, Βοσνία Ζεγουβίνη, θα καταθέσω μία ή δύο τροπολογίες αύριο. Θα ήθελα όμως να χωριστεί σε δύο παραγράφους. Η πρώτη παράγραφος θα λέει ότι χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη τελικά σημειώνει πρόοδο στην επίτευξη του οδικού χάρτη που έχει μπροστά της. Και στη δεύτερη παράγραφο θα ήθελα να γίνει μια τροποποίηση. Θα ήθελα να αναφερθεί ότι σημειώνουμε ότι η Διεθνή κοινωνία έδρασε ευτυχώς στη Βοσνία Ζεγοβίνη αλλά ότι ελπίζαμε ότι όταν η Διεθνή κοινωνία δρά εκεί δρά βάσει των συμφωνιών που ήδη υπάρχει μεταξύ των ε, συμβαλωμένων μελών. Δεν έκανε τη συζήτηση με βάση αυτών των συμφωνιών και γι' αυτό πέτυχε. Έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία και θα θέλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι είναι σωστό το σημείο 15 ε, για την Αλβανία και το Μαυροβούρι να τα αναφέρουμε από κοινού. Θα υπάρχουν θέματα που πρέπει να αναφέρουμε ξεχωριστά για την Αλβανία γιατί στην ε, Αλβανία η αντιπολίτευση βγαίνει στο δρόμο αντί να βγει στη Βουλή. Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση από την ε, δημοκρατική, το Δημοκρατικό Κόμμα και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση είναι αυτό ήδη απόδειξη οριμότητας. Δεν θα το φανταζόταν κανένας. Αυτό θα πρέπει να το χαιρετήσουμε και θα πρέπει να καλέσουμε την αντιπολίτευση να αναλάβει το έργο της επιτέλους. Πρέπει να μπει στη Βουλή, όχι στο δρόμο. Και έχω να πω ότι εδώ στο σώμα πολλές φορές είχα ψηφίσματα που αναφερόμουν στην τότε αντιπολίτευση που σύμπανε στην κυβέρνηση και την καλούσα να πάει στη Βουλή και να πάψει να κατεβαίνει μόνο στους δρόμους. Και γι' αυτό δεν πρέπει τώρα να μην υπενθυμίσουμε στη σημερινή αντιπολίτευση ότι έχει εκλεγεί για να εργάζεται στη Βουλή. Για αυτά τα σημεία λοιπόν θα υποβάλω αύριο τροπολογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Πάκ, ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά σας. Η συνάδελφος Όμεν Ρόιτεν είναι στη θέση της. Ε, ήθελα βέβαια να της δώσω το λόγο για πρώτη, διότι ήταν η συγγήτρια για την Τουρκία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορώ να είμαι σύντομη, διότι αύριο θα μιλήσουμε για την έκθεση πρόοδου. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό να αναφέρει κανείς κάποια σημεία όσον αφορά στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και την έκθεση πρόοδου. Το κράτος δικαίου είναι πολύ σημαντικό για την Τουρκία και υπάρχουν κάποια, επίσης και κάποια διμερεί θέματα τα οποία θα ήθελα να περιλαμβάνονται στο ψήφισμα. Στην παράγραφο για την Τουρκία λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, στη δικαιοσύνη. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα στην Τουρκία. Διότι δεν υπάρχει σωστή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ακόμα αυτό, ε, εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλο πεδίο ε, μεταρρύθμισης. Πρέπει να υπάρξει όμως συνένεση στην ε, Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, να υπάρχει ομοφωνία. Ένα άλλο ζήτημα είναι η Κύπρος. Την περασμένη εβδομάδα όλοι οι συνάδελφοι μιλούσαν για τα προβλήματα σχετικά με την Κύπρο. Υπάρχει η Συμφωνία της Άγκυρας, υπάρχει μια συμβατική ρύθμιση με την Τουρκία. Γνωρίζω βέβαια ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν ξέρω ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πούμε κάτι και από αυτού και τελευταίο σημείο. Κατά την ε, περασμένη εβδομάδα ασκήθηκε ε, μεγάλη κριτική στα όσα είπε ο κύριος Ερντογάν στο Ιράν. Δήλωσε ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι με το Ιράν, αλλά ε, εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ζήτημα να είμαστε καλοί φίλοι, δεν αρκεί να είμαστε καλοί φίλοι. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να ξέρουμε πώς βλέπει το πυρηνικό ζήτημα, το ζήτημα των πυρηνικών όπλων ε, στο Ιράν. Το άνοιγμα προς τους Κούρδους, το δημοκρατικό άνοιγμα προς τους Κούρδους είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και πρέπει να το επισημάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά σχετικά με την έκθεση Τουρκίας. Η κυρία Νέιτς που είναι συντονίστρια της ομάδας της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την εξαίρεση που κάνατε υπέρ μου, δηλαδή να μην μιλήσουν μόνο βουλευτές του ΕΛΚ. Λέει ο Μιλήτρια. Χαίρομαι Ιδιαίτερα για το κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε και τροπολογίες θα κατατεθούν αύριο. Για το σημείο 3 έχω μπροστά μου το κείμενο στα αγγλικά. Στο σημείο 3 καλούνται όλοι οι χώρες να κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεπεράσουν τις διαφωνίες και τα προβλήματα που έχουν με τους γειτόνους τους. Λέγεται όμως επίσης ότι θα πρέπει να λυθούν διμερώς τα προβλήματα, τους ενδιαφερόμενους. Και οι διμερείς διαφορές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο για τις χώρες ε, στην κατεύθυνσή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Νομίζω λοιπόν ότι εδώ το σπρώχνουμε αρκετά το πράγμα. Εμείς ήδη έχουμε εμπειρίες ε, με χώρες ε, στις οποίες ε, αφήσαμε να γίνουν μέλη πριν λύσουν τα υπάρχοντα προβλήματα. Και αυτές οι χώρες τα σέρνουν μαζί τους αυτά τα προβλήματα χωρίς να γίνεται ποτέ νήξη για μια οποιαδήποτε πραγματική λύση. Πρέπει λοιπόν εδώ να αλλάξουμε την διατύπωση αυτή που θεωρώ ότι είναι πολύ γενναιόδορη. Για την Κροατία εγώ πιστεύω και είμαι πάρα πολύ ειλικρινής ότι η Κροατία κατάφερε να προχωρήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να κλείνει τις διαπραγματεύσεις μέχρι το 2010. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο είναι λογικό εδώ να το λέμε τόσο καθαρά πια το θέμα διότι θα μπορούσαμε απλώς να περιοριστούμε να εκφράζουμε την ευχή δηλαδή να λέμε ελπίζουμε ότι η Κροατία θα ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις στο αργότερο μέχρι το 2010 Πιστεύω όμως ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι γιατί δεν ξέρουμε τελικά πώς θα καταλήξουν αυτές οι διαπραγματεύσεις τώρα για την Τουρκία. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν μιλάω εξ ονόματος της ομάδας μου εδώ, μιλάω προσωπικά. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια τεράστια παρεξήγηση με την Τουρκία. Από τη μια λέμε στην Τουρκία τι πρέπει να κάνει για να βελτιώσει την κατάσταση και συμφωνώ με αυτό, αλλά ταυτόχρονα εμείς ε, καλούμε την, τουρκική κυβέρνηση να συντονίζει την εξωτερική της πολιτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα νομίζω ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ή έχουμε ένα διάλογο μεταξύ ίσων και μπορούμε να καλούμε μια χώρα να καταλήγει σε, να, να ασκεί εναρμονισμένη πολιτική με, με την δική μας εξωτερική πολιτική ή αλλιώ τους λέμε, κοιτάστε θα κάνετε αυτό, αυτό και αυτό, λείπει το τάδε το τάδε ζητούμενο και δεν ε, θα τους καλούμε να ασκούνε ε, ομόλογη εξωτερική πολιτική. Τώρα για το Κυπριακό πιστεύω ότι οι ευχές ε, θα πρέπει να εκφράζονται και για τα δύο μέρη αν θέλουμε να προχωρήσει η κατάσταση. Αυτές ήταν οι αρχικές μου παρατηρήσεις και όπως σας είπα θα παρουσιάσω και τις σχετικές τροπολογίες. Και για να ολοκληρώνω πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με την ε, κυρία Πάκα ε, σχετικά με τις ε, διευκολύνσεις για τις θεωρήσεις, δηλαδή τις βίζες με τη Βοσνία, Ζεγοβίνη και το Κόσοβο. Όπως έλεγε και η Σάρα Λότφορντ πρέπει να έχουμε μία νέα αντιμετώπιση διότι ορισμένοι σίγουρα θα ολοκληρώσουν την πορεία τους νωρίτερα από τους άλλους αλλά αν βρούμε κι εμείς μία διατύπωση που να αντικατοπτρίζει αυτή την κοινή θέση θα την υποστηρίξω με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ κυρία Νέιτς. Δεν υπάρχει εξαίρεση προσωπική προς εμάς, Κυρία Νέιτς, ε, πρόκειται για εξαίρεση προς όλους ε, τους συναδέλφους από όλα τα κόμματα. ο κύριος Ντίγκενινγκ, συντονιστής της ομάδας του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι καλή έκθεση. Δεν έχουμε βασικές αντιρρήσεις. Και εκπονήθηκε ε, στο πλαίσιο καλής συνεργασίας μεταξύ των συγγητών. Δεν είναι μια έκθεση για, γενικότερα για τη στρατηγική, αλλά αφορά τα Βαλκάνια, την Ισλανδία και την Τουρκία. Αλλά παρόλα αυτά είναι χρήσιμο να αναφέρει κανείς κάποια βασικά θέματα και κάποιες εξελίξεις. Επί σειράν ετών, οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τις εκρεμείς θεσμικές μεταρρυθμίσεις ως πρόφαση ε, για να καθυστερήσουν την ε, διαδικασία. Τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμη να συνεχίσει, να προχωρήσει ε, στο ζήτημα της διεύρυνσης. Τώρα, το θέμα της ε, απελευθέρωσης ε, του μηχανισμού χορηγήσης δια... θεωρήσεων, κατάργηση δηλαδή θεώρησης διαβατηρίων. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε και να οικοδομήσουμε πάνω σε όσα έχουμε ήδη επιτύχει στην Επιτροπή μας. Αν είναι απαραίτητο, ας επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τις θέσεις μας. Χρειάζεται κάποια αναδιάταξη σε κάποια σημεία. Ίσως πρέπει να τονίσουμε ή να προσθέσουμε στις παραγράφους όπου μιλούμε για την περιφερειακή συνεργασία να αναφέρουμε την ανάγκη για απελευθέρωση του εμπορίου γιατί αρκετές χώρες βρίσκονται ακόμα πολύ πίσω. Στο έγγραφο στρατηγικής της Κομισιόν ένα σημείο που θεωρώ σημαντικό και ίσως πρέπει να περιληφθεί στο ψήφισμά μας είναι η ανάγκη να φέρουμε τους πολίτες αυτών των χωρών και τις κυβερνήσεις τους ή και τι διοικήσει του πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πολιτική ενημέρωση και ειδικά μέτρα ώστε να έρθουν και οι πολίτες πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην είναι απλώς μια διοικητική προσπάθεια, μια προσπάθεια του κράτους, αλλά να μπορέσουν και οι πολίτες να έχουν αυτό το διάλογο με τα θεσμικά μας όργανα. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Η κυρία Ντόρις Πακ μάλλον φεύγει. Ε, για την Αλβανία ήθελα να πω. Συμφωνώ μαζί της ότι δεν είναι καλό να βάζουμε την Αλβανία και το Μαυροβούνιο μαζί σε μία παράγραφο, σε ένα σημείο. Αλλά Δεν μπορούμε ουσιαστικά να μιλάμε για καλό πολιτικό περιβάλλον στην Αλβανία και καλή λειτουργία της διοίκησης και της κυβέρνησης όταν σχεδόν το ίμιση των μελών του Κοινοβουλίου δεν συμμετέχουν στο έργο, στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε έκκληση, αλλά πρέπει να, μια, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αν αυτή είναι εκτός, έχουν τους λόγους τους να είναι εκτός. Ίσως η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό και να κοιτάξουμε, να εξετάσουμε την κατάσταση από πιο, πολύ πιο κοντά. Δεν νομίζω ότι σε μια χώρα η οποία επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η, η αντιπολίτευση θα θέλει να μένει εκτός. Ε, εδώ υπάρχει μια αντίφαση την οποία πρέπει να βάλουμε υπόψη. Ο κύριος Στάλερ, εισηγητής για τη Μακεδονία, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στην σημασία της έκθεσης και της, ε, του ψηφίσματος. Είναι γενικά μια καλή έκθεση και θα πρέπει πριν από το Δεκέμβρη να αποστείλουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Η περιοχή του Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμιά φορά όμως δίνουμε την εντύπωση ότι έχουμε κάπως κουραστεί να ασχολούμεθα με την περιοχή αυτή. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τη Μέση Ανατολή, με το Αφγανιστάν, με τις κλαμολογικές ε, ε, κρίσεις κλπ. Αλλά θα πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα εδώ, στην αυλή μας. ε, βασίζομαι και στη νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και το έχει αμελήσει αυτό το τελευταίο καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, θα είναι σοβαρός παράγοντας ε, ισχύω χωρίς την ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Ό,τι και αν σκεφτόμαστε για τα Δυτικά Βαλκάνια, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους φέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να ζούμε με τις αυταπάτες ότι μπορούμε να απομονώσουμε την περιοχή αυτή. Χωρίς αυτές τις ε, χώρες δεν μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί και υποκοδομητικοί ως Ένωση. Και γι' αυτό νομίζω ότι και η χρονική στιγμή του ψηφίσματος και το περιεχόμενο είναι πολύ καλό. Μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο αν χρειάζεται, αλλά δεν θα χρειάζεται νομίζω να περιμένουμε μέχρι τα ε, Χριστούγεννα. Για την ε, τέως Υπουργική ε, Δημοκρατία της Δημοκρατίας νομίζω το κείμενο είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης το θέμα του Κωσυφοπεδίου θα πρέπει να το αναφέρουμε πιο αναλυτικά. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επιληθούν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην Πρίσινα και στα Σκόπια. Έχουν βρεθεί καλές λύσεις και μας έχουν αποδείξει πώς μπορούν να επιληθούν προβλήματα σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Τάλερ. Αυτή η πρώτη φάση των τοποθετήσεων είχε να κάνει με τους εισηγητές και τους συντονιστές και δεν περιόρισα το χρόνο μιλίες. Όμως ε, η ώρα ε, με υποχρεώνει να περιορίσω το χρόνο ομιλία. Οπότε οι αναπληρωτές δεν μιλάνε. Κυρία Γιαννάκου, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ ε, για το ψήφισμα αυτό. Έχω ορισμένε παρατηρήσεις να κάνω ε, και, και θα κάνω κάποιες τροπολογίες αύριο. Οι παρατηρήσεις αυτές ε, κυρίως αφορούν ε, στο 9 και 10, δηλαδή στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ε, θέλω να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα στη χώρα, πλην ενός το οποίο είναι πολύ μικρό προς τα δεξιά, ε, έχουν κάνει την τοποθέτησή τους, δέχονται μία σύνθετη ονομασία και πρέπει να τηρηθούν όσα προβλέπονται από τα Ηνωμένα Έθνη, να συμφωνήσουν δύο χώρες δηλαδή, ε, σε ένα όνομα. Επομένως η Ελλάδα έχει κάνει τις κινήσεις που πρέπει και δεν υπάρχει περίπτωση ε, η νέα κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό δηλαδή ε, που γράφετε εσείς εδώ πέρα. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να, και δεν θέλει να εμποδίσει το δρόμο της χώρας αυτής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τηρήσει τα υπεσχημένα και τους κανόνες και από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων χωρών ε, δεν πρέπει να, θεωρείται ότι είναι ευθύνη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να κάνουν όλες τις υποχωρήσεις που χρειάζονται προκειμένου να ενταχθούν νέες χώρες και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διακρίνεται και από αλληλεγγύη και από αλληλοβοήθεια και από στήριξη μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό και θα υποβάλω τροπολογίες κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου. Για δύο λεπτά η κυρία Εμπρίζα Ζήτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα είπε η κυρία Πακ. Θα ήθελα όμως να με επιτρέψετε να προσθέσω και κάποια σημεία και να υποβάλω και μία τροπολογία. Υπάρχουν κάποια σημεία που αφορούν όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Παραδείγματος κάνει κατά πολέμηση οργανωμένων κλίματος, διαφθορά, συνεργασία με το Διεθνές ε, ε, Ποινικό Δικαστήριο κλπ. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι πολύ θετικά. Παραδείγματο χάρη συνεργασία με το ποινικό δικαστήριο. Ναι. Αλλά Ε, αναφέρονται και κάποιες, ε, θα μπορούσαν να αναφερθούν κάποιες ε, χώρες ρητά. Το θέμα της διαφθοράς επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί. Αλλιώς δεν είμαστε συνοπείς και αυτό δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Και θα πρέπει εδώ να προειδοποιήσουμε και η Σερβία που έχει επίσης προβλήματα. Θα υποβάλουμε λοιπόν κάποιες σχετικές ε, τροπολογίες. Για τη Βοσνία μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Πακ ότι το κείμενο εν μέρη δεν είναι πάρα πολύ επιτυχές. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία που είναι θετικά και μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Πακ. Αλλά σας είπα θα υποβάλω και κάποια τροπολογία και εδώ. Ευχαριστώ κυρία Ζίτ. Η κυρία Κόβατσεφ για δύο λεπτά. Ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Συζητούμε τώρα το σχέδιο ψηφίσματος ε, επί του ε, κειμένου της στρατηγικής της διεύρυνσης και βέβαια κάθε ένα από τα σημεία του ψηφίσματος θα τα συζητήσουμε αύριο. Και δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτού του σχεδίου ψηφίσματος και των απόψεών μας για, τα επιμέρου για τις επιμέρους χώρες αργότερα. Στο σημείο 9 παραδείγματο χάρη για τη Μακεδονία λέει να καθοριστεί η ημερομηνία για την έναξη των διαπραγματεύσεων. Ενώ στην έκθεση της κυρίας Στάρα ε, λέμε ότι αναμένει ε, την έναρξη διαπραγματεύσεων στο άμεσο μέλλον. Εδώ πρέπει να υπάρξει διόρθωση. Στην τελευταία εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη Μακεδονία, αναφερθήκαμε στα προβλήματα στα προβλήματα ε, που υπάρχουν μεταξύ της χώρας αυτής και των γειτονικών χωρών για το περιεχόμενο των βιβλίων ιστορίας για, τους, για τις επαιτίους ε, εορτασμού ιστορικών γεγονότων δεν θα πρέπει αυτά να εμπλέκονται στην επίλυση των πολιτικών ζητημάτων και οι αρχές της Μακεδονίας θα πρέπει να εγγυηθούν και τα δικαιώματα εκείνων ε, ε, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως ε, επίσημοι ως ανήκοντες επίσημα σε κάποια από τις μειονότητες. Η κυρία Κοπά. Δύο λεπτά. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το κείμενο το οποίο έχετε υποβάλει και για την προσπάθειά σας να κρατηθεί και να ενισχυθεί η δυναμική της διεύρυνσης η οποία το τελευταίο καιρό βάλετε πάρα πολύ ευρωπαϊκά ε, κυρίως σε ό,τι αφορά την Τουρκία όπου έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια ότι έχει επιχειρηθεί ακόμα και η λέξη ένταξη να μην υπάρχει στα κείμενα αλλά ακόμα και για την περίπτωση των ε, Δυτικών Βαλκανίων όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να βγει ένα κείμενο το οποίο να δείχνει την ε, θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσει η Ευρώπη σε αυτή τη διαδικασία. Ε, θέλω να κάνω μερικά πολύ σύντομα σημεία. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της Σερβίας. Ε, το κείμενο πράγματι αναγνωρίζει την πρόοδο, αναγνωρίζει τη μονομερή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας. εγώ θα επιθυμούσα να υπάρχει και μία αναφορά στην τελευταία δήλωση του κύριου Μπράμερτς για το πόσο έχει προχωρήσει η Σερβία στο θέμα του δικαστηρίου, του ICTY, ε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, ακόμα και για να αναγραφεί στα συμπεράσματα το θέμα της ε, ε, μονομερούς εφαρμογής, οπότε το να αναγραφεί αυτό το θετικό για τη Σερβία έχει μεγάλη σημασία. Δεύτερο σημείο έχω, το έχω ξαναπεί ότι ανεξάρτητα και αν στα κείμενα βάζουμε ότι τα διμερεί θέματα δεν έχουν σημασία και δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην διεύρυνση και στην ένταξη αυτό είναι μια πραγματικότητα. το θέμα είναι πώς μπορούμε τα εναπομείναντα τα ζητήματα των βαλκανίων να τα λύσουμε μέσα σε μια ενταξιακή δυναμική δηλαδή να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε διατηρώντας ανοιχτό το στόχο της διεύρυνσης και αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Στο θέμα της Τουρκίας, ε, εγώ συμφωνώ με την ε, κυρία Ούμεν Ρόιτεν ότι ε, πρέπει να γίνει όλη η συμπλήρωση και να αναφερθούν τα σημεία που λέει. Θα ήθελα όμως να γίνει σαφής αναφορά για το θέμα καλής γειτονίας παρά τα θέματα που έχει βελτιώσει η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα έχει εμφανιστεί κλιμάκωση σε στρατιωτικό επίπεδο στο Αιγαίο το οποίο είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος οδηγός για μια υποψήφια χώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια για την Ισλανδία, για το σημείο 16. Καταρχήν, να, σημειώσω, να τονίσω κάτι σχετικά με τις Ισλανδικές αρχές οι οποίες ε, πολύ γρήγορα, δηλαδή σε ένα μήνα και λίγες μέρες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που έστησε η Κομισιόν. Το είδαμε αυτό δηλαδή και με τον κύριο Γιώχανσον που είναι και ο πρέσβης της Ισλανδίας ε, παρά τη ενώση και είναι και ο αρχηγός των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Γιώχανσον λοιπόν είπε και ξέφρασε την επιθυμία ότι η Κομισιόν πρέπει να απαντήσει γρήγορα στο ερωτηματολόγιο που έστειλαν οι Ισλανδοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο τεράστιος διχασμός της κοινή γνώμης για το ένταξη ναι, ένταξη όχι, αυτό και τα κόμματα της, ε, του συνασπισμού της κυβέρνησης διαφωνούν μεταξύ τους. Το είδαμε αυτό και όταν είχαμε εδώ τα μέλη ε, του Ισλανδικού Κοινοβουλίου στην αντιπροσωπεία. Εγώ λοιπόν θα καταθέσω μία τροπολογία σχετικά. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Δύο λεπτά. Ο κύριος Μαυρονικόλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο κείμενο σε ό,τι αφορά την Τουρκία και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, στην αναφορά του κειμένου για το κυπριακό πρόβλημα. Πιστεύω ότι το κείμενο δεν είναι αρκούντος ικανοποιητικό στην αναφορά του για ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία όχι μόνο δεν έχει υλοποιήσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας δεν έχει αναγνωρίσει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν έχει ανοίξει τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και το εμπόριο μέχρι αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, δεν έχει συμβάλει καθόλου στις συνομιλίες που γίνονται στο νησί, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση επαναληπτικά μιλά για λύση μεταξύ δύο κρατών. Άρα θα υποβάλουμε τροποποιήσεις ούτως ώστε το κείμενο αυτό να είναι αρκούντος ενισχυτικό για ένα πρόβλημα που αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η σημερινή διακυβέρνηση έχει διαφυλάξει τις απόψεις και θέσεις της για τον Δεκέμβριο με την πιθανότητα να υποβάλουμε κυρώσεις για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Άρα θεωρώ ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη κύριε Πρόεδρε ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι και πρόβλημα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. για δύο ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας πω ποιες είναι οι ανησυχίες μου βάζουμε διάφορες χώρες σε ένα ψήφισμα. Πολλές χώρες, διαφορετικές χώρες, σε μερικές περιπτώσεις πάρα πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Νομίζω λοιπόν ότι το έγγραφο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά ισορροπημένο και θα πρέπει να έχει πολύ λεπτές ισορροπίες. Νομίζω ότι ε, έχει ε, κάποια ισορροπία. Με κάποιες τροπολογίες από την Doris Πακ και κάποιους άλλους, αυτή η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί. Ωστόσο, πρέπει ε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για κάθε χώρα, δεν νομίζω ότι θα επιτύχουμε το ε, επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι θα δοθεί περισσότερη έμφαση σε κάθε χώρα, ενώ το έγγραφο αυτό θα πρέπει να είναι ένα πολύ συνεκτικό και καθαρό έγγραφο. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν να επιδείξετε ηγετική ικανότητα ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η ισορροπία, η λεπτή εσωτερική ισορροπία στο έγγραφο. Ευχαριστώ. Θα το πω στο τέλος, βέβαια το προδικάζω τώρα, θα τα πω και στην αρχή προσπάθησα να αφήσω όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο στη δική σας γνώμη. Ο κύριος Κασουλίδης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο επί ενός σχολείου της κυρίας Νέιτς η οποία είπε ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αμφότερες τις πλευρές στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Το ερώτημα είναι ποιες είναι οι πλευρές. Διότι εάν σύμφωνα με κάποιους και ιδιαίτερως ε, σύμφωνα με την Τουρκία οι δύο πλευρές είναι οι δύο κοινότητες της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Τουρκία για τις δικές της υποχρεώσεις που είναι μια υποψήφια χώρα εκτός Κύπρου και από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ίδιο το κεφάλαιο περί ασφάλειας κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. Και τώρα θα περάσουμε στους αναπληρωτές. Ο κύριος Πένσιν για δύο λεπτά έχει τον λόγο. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ ε, δύο σχόλια Νομίζω πραγματικά ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναφερθούμε σε θέματα συγκεκριμένα. Μειονότητες, παραδείγματος χάρη στην Τουρκία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του Οικονομικού Πατριαρχείου και της κυβέρνησης ε, της Τουρκίας. Υπάρχουν ε, οι σχολές ε, των ιερωμένων που έχουν κλείσει, υπήρξε κάποιος διάλογος σχετικά, αλλά λέγεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κοινότητες. Ποιες χριστιανικές ομάδες πλήττουν εδώ από αυτή την κυβέρνηση και τι πρέπει ακριβώς να εξεταστεί. Κατόπιν, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ το θέμα της Τουρκίας και να σας πω ότι θα πρέπει ακριβώς να πούμε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, <clears throat> όταν στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, λέω ποια είναι τα επίμαχα σημεία. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις για να μπορέσει κάποια στιγμή να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σφέντσον. Το λόγο έχει στον Αλβό Βάιγκελ, που είναι συγκεκριτή την Κροατία. Ε, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την έκθεσή σας που είναι σύντομη μεν αλλά πολύ πλήρης. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το κείμενο δεν θα πρέπει να κατακαιρματιστεί. Λίγα σχόλια. Συμφωνώ με την παρατήρηση ότι το σημείο 3 θα πρέπει να διατυπωθεί κάπως πιο προσεκτικά. Ούτως ώστε διμερεί ανοιχτά θέματα να λέμε λέω ότι τα ανοιχτά θέματα θα πρέπει να επιληθούν από τα δύο ενδιαφερόμενα μέλη. Όταν πρόκειται όμως για θέματα σύνορων θα μπορούσε να είναι το θέμα πιο σημαντικό και γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να υποβάλω μία νέα διατύπωση αύριο και επίσης όταν αναφερόμαστε στο κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να αναφερθούμε στο ότι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση του κοσυφοπαιδίου για την προστασία της σερβικής μειονότητας γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σχέση με τη γειτονική χώρα τη Σερβία και θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι οι Σέρβοι στο κοσυφοπαίδιο δεν αισθάνονται ακόμα επαρκώς προστατευόμενοι και ασφαλείς. Και τέλος θα ήθελα να προτείνω η Αλβανία και το Μαυροβούνι να αναφερθούν σε δύο διαφορετικές παράγραφοι σαν δύο χώρες. Να μην τις συνενώνουμε σε μία παράγραφο. Και να αναφερθούμε σε ό,τι έχει κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά. Ε, ευχαριστώ. Έχουμε ένα πρόβλημα με τους διερμηνείς. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Κουμουτσάκο αν θα μπορούσε να είναι συντομότερος των δύο λεπτών διότι θέλω να ακούσω και την Κομισιόν και θα περιορίσω στο ελάχιστο την δική μου απάντηση. Κύριε Κουμουτσάκο, σύντομα παρακαλώ. Λιγότερο από δύο λεπτά αν τα καταφέρετε. Ήταν εσείς τόσο αναλυτικός που μου πείσατε ότι πρέπει να είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Ευχαριστούμε για το κείμενο που καταθέτετε πιστεύω σταθερά και στεναρά στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη πρέπει να εκπληρώνουν πλήρως τα σχετικά κριτήρια και τα προαπαιτούμενα. Στο πλαίσιο αυτό έχει εξαιρετική σημασία ο σεβασμός της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας. Ειδικά για τα Δυτικά Βαλκάνια αυτό είναι θέμα πρώτης προτεραιότητος Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω και συμφωνώ εδώ με την κυρία Κοπάλα και με άλλους που μίλησαν ότι δεν μπορούμε να προσποιούμεθα ότι τα υπάρχοντα προβλήματα σχέσεων καλής γειτονίας δεν επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πορεία των ενδιαφερομένων για ένταξη χωρών. Αυτή είναι μια γενική θέση που έχει επίπτωση και σε μια σειρά άρθρων του ψηφίσματος που πρόκειται να συζητήσουμε αύριο. Γι' αυτό και θα κατατεθούν σχετικές τροπολογίες ε, στα άρθρα κυρίως 3, 9, 10 αλλά και 11. Είναι μια βασική αρχή ο σεβασμός των ε, σχέσεων καλής γειτονίας που δεν μπορούμε να προσποιούμε ότι δεν επηρεάζει την ενταξική πορεία των ενδιαφερομένων χωρών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Το λόγο έχει η Επιτροπή ο Δόκτωρ Τιμοσούμα. Παρακαλώ σύντομα έχουν πρόβλημα οι διερμηνείς για τα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη για το ψήφισμα, που, ψήφισμα το οποίο είναι σύμφωνο με τα συμπεράσματα της Κομισιόν. Κάποια σχόλια μόνο επί κάποιων σημείων και οι προτάσεις θα δοθούν μετά στη Γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημείο 2. Διεθνές Δικαστήριο θέση του Συμβουλίου είναι ότι η πλήρη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία είναι θεμελιώδης σημασία. Σημείο 10. Φιρόμ, Πουγδουμού. Θα είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι η επίλυση του ζητήματος του ονόματος είναι θεμελιώδου σημασίας για να αρθεί αυτό το εμπόδιο προς την κατεύθυνση της εσωμάτωσης της χώρας αυτής. Σημείο 11. Η Τουρκία θα πρέπει να εκπληρώσει απολύτως τα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγης. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το άρθρο 301 στο ε, ποινικό κώδικα δεν χρησιμοποιείται συστηματικά πλέον για την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα αυτή. Και υπάρχει μια αυξανόμενη ε, ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση στην τουρκική κοινωνία για θέματα τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα. Σύμφωνα με τον νόμο του 2000 σχετικά με τα ιδρύματα και τα δικαιώματά τους και ο διάλογος το που έχει ανοίξει η κυβέρνηση με τους Αλεβίτες και τις μη μουσουλμανικές ε, κοινότητες εφαρμόζεται ομαλά. Ωστόσο θα πρέπει κανείς να σημειώσει ότι ο νόμος για την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της θρησκείας, ο νόμος αυτός δεν είναι δεν προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις ε, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως προς το ε, θέμα της ε, Αλβανίας, η Αλβανία θα πρέπει να προσαρμοστεί προς τις απαιτήσεις που έχουμε ε, επιβάλλει. Σημείο 16. Η έκθεση αναφέρει το υψηλό επίπεδο ευθυγράμμιση τη Ισλανδία με το κοινοτικό κεκτημένο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα γενικότερα κριτήρια τη Κοπενχάγη, θα μπορούσε κανεί να αναφέρει την ε, καθιερωμένη, εδρεωμένη δημοκρατική παράδοση της χώρας αυτής. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για τις συντομίες σας. Δεν εγκομιάζω. Θα κοιτάξω να είμαι και εγώ εξίσου σύντομος. Σημείωσα λοιπόν τις τοποθετήσεις σας, κριτικά σημεία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, διάκριση μεταξύ των δύο, συμμετοχή αμφωτέρων, η Τουρκία, με όλες τις, τις πολυπλοκότητες, Φυρόμ, Μακεδονία. Υπάρχουν επίσης ε, θέματα σεναρίων, ε, εμπορική απολευθέρωση, συνεργασία της Σερβίας με το δικαστήριο της Χάγης, τέλος πάντων, απλούστευση όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω όλα αυτά με ε, την απόλυτη διαθεσιμότητά μου να συνεργαστώ με όλους σας. Οι τροπολογίες λοιπόν μέχρι